Πρόκειται συγκεκριμένα για την έκθεση Vivian Ρέντινγκ για τις διαπραγματεύσεις επί της Συμφωνίας της Συναλλαγής των των Υπηρεσιών. Κυρία Ρέντινγκ, έχετε το λόγο. Euh, κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, ενώ ε, από το 2013 διαπραγματευόμαστε με 23 χώρες, το 70% δηλαδή του εμπορίου υπηρεσιών, η ΤΙΣΑ ε, παραμένει άγνωστη ε, στο ευρύ κοινό. Ωστόσο, σύντομα θα υποκείμεθα στους κανόνες αυτής της συμφωνίας. Όταν τηλεφωνούμε, όταν χρησιμοποιούμε την πιστοτική μας κάρτα, όταν παίρνουμε τις συγκοινωνίες ε, σε κάποια χώρα του εξωτερικού, όταν ε, συνδεόμαστε ηλεκτρονικά σε κάποια ιστοσελίδα για να ψωνίσουμε κάτι ε, ή σε κάποιο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, σε χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, κανείς δεν θα μείνει εκτός και άρα πρέπει να γνωρίσουμε τις διατάξεις αυτής της συμφωνίας. Η Κομισιόν διαπραγματεύεται εξ ονόματος της Ένωσης, το Κοινοβούλιο όμως το οποίο ελέγχει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα χαράξει πολύ σαφή κατευθυντικές κατευθυντήριες γραμμέ. Όπως λοιπόν μαρτυρεί και η έκθεση, τη οποία θα αποφανθεί την Τετάρτη το σώμα, είναι τέτοιες οι προκλήσεις που οι ευρωβουλευτές συμπαρατάσσονται ξεχνώντας ε, τις πολιτικές τους διαφορές ε, για να ε, αλλάξουν τον προσανατολισμό της κοινής εμπορικής πολιτικής της Ένωσης και σε ό,τι αφορά την ουσία και σε ό,τι αφορά τη μορφή των διαπραγματεύσεων. Σε ό,τι αφορά καταρχάς τη μορφή των διαπραγματεύσεων, πρόκειται για πραγματική τομή γιατί διαμακρώνει οι διαπραγματεύσεις γίνονταν και κλεισμένων των θυρών μετά στις εκλογές του 2014 αλλάζει η κατάσταση. Οι βασικές ε, πολιτικές ομάδες ε, παρακολουθούν ε, αδιάλειπτα κάθε γύρο διαπραγματεύσεων ενώ υπάρχει και έντονο εσωτερικός διάλογος εντός κοινοβουλίου με την διαβούλευση με οκτώ κοινοβουλευτικές επιτροπές αλλά και εκτός θεσμικών οργάνων να υπάρχει διαβούλευση με την κοινωνία των πολιτών κυρίως. Κατόπιν δικού μας αιτήματο η εντολή ε, του Συμβουλίου και οι προτάσεις ε, του Κοινοβουλίου δημοσιοποιήθηκαν ήδη και θέλω να σας ευχαριστήσω κυρία Επίτροπε διότι και εσείς ε, βοηθήσατε προς αυτή την κατεύθυνση. Με την έκθεση μας θέλουμε να προχωρήσουμε ακόμη περισσότερο, να έχουμε περισσότερη διαφάνεια. Έρχομαι τώρα στην ουσία. Και εδώ βλέπουμε ριζικές αλλαγές ως ε, βουλευτές, ως αιρετοί ε, έχουμε την ευθύνη να καθορίζουμε ε, την τίζα που θέλουμε και την τίζα που δεν θέλουμε. Το δικό μας μήνυμα είναι σαφές. Θέλουμε καλύτερη διεθνή ρύθμιση και κανονισμούς δίκαιους και στέρεους. Πιο συγκεκριμένα, στην έκθεση αυτή υπάρχουν κάποιες ε, γαλάζιες γραμμές, περισσότερα αμοιβαιότητα με τις εξωτερικές αγορές, ιδίως στους τομείς των τηλεπικοινωνιών, των μεταφορών και των δημοσίων ε, συμβάσεων. Περισσότερα δικαιώματα για τους καταναλωτές κατά καταχρήσεων, όπως είναι τα τέλη περιαγωγής ή το spam. Περισσότερα επίσης ωφέλη και πλονεκτήματα για τις μικρομεσαίες επιχείρησεις και τέλος περισσότεροι συμμετέχοντες στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων όπου θα μπορούσαμε να φανταστούμε να κάθεται και η Κίνα. Ποιε είναι τώρα οι κόκκινε γραμμέ, πολύ άριθμε και αυτέ. Δεν θα πρέπει, μάλλον οι τηλεπικοινωνικέ υπηρεσίε, θα πρέπει να ε, εξαιρούνται και θα πρέπει τα δικαιώματα, τα θεμελιώδη, δηλαδή η προστασία δεδομένων να διασφαλίζονται, η ε, διακίνηση των προσώπων να περιορίζεται στην προσωρινή διακίνηση ε, προσοντούχων ανθρώπων στο πλαίσιο σύμβασης. Τέλος, ε, σε ό,τι αφορά επιθετικά και αμυντικά μέτρα. Αυτά είναι αδιαίρετα και δεν μπορεί να υπάρξει συμφωνία χωρίς προστασία. Αλλά και ούτε και προστασία χωρίς συμφωνία μπορεί να υπάρξει. Το 25% των παγκόσμιων εξαγωγών και το εμπορικό πλεόνασμα των 160 δις Νομίζω ότι με αυτά τα στοιχεία μπορούμε να αλλάξουμε τα δεδομένα ε, με κανόνες πιο δίκαιους και πιο σταθερούς. Την Τετάρτη, αγαπητοί συνάδελφοι, θα έχετε τη δυνατότητα να εκπέμψετε ένα ηχηρό μήνυμα προς τους διαπραγματευτές, έτσι ώστε οι διαπραγματεύσεις να στραφούν προς τη σωστή κατεύθυνση, προς όφελος των επιχειρήσεών μας, προς όφελος ε, των Ευρωπαίων πολιτών. Ψηφίστε λοιπόν κατά της έκθεσης, τι θα, τι θα πει, ψηφίστε κατά του ε, καθεστώτος, ε, κατά της αμοιβότητας και κατά ε, των κανόνων. Αν ψηφίστε υπέρ όμως έκθεσης, τι θα πει, θα πει αλλαγή, θα πει διαφάνεια, προάσπιση των αξιών μας, των συμφερόντων μας. Άρα να ψηφίσετε υπέρ γιατί αυτό σημαίνει ότι η Κομισιόν δεσμεύεται με ένα σαφές κοινοβουλευτικό, με μια σαφή κοινοβουλευτική εντολή. Πρέπει λοιπόν να αναλάβουμε τις ευθύνες μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Η Επίτροπος Μάστρομ έχει το λόγο. Uh, Ευχαριστώ και καλό απόγευμα. Η Επιτροπή θα ήθελε να ευχαριστήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τη μεγάλη εμπλοκή του για το γεγονό ότι έχει συζητηθεί το ζήτημα σε τόσε πολλέ επιτροπέ και επίση για το έργο σα, κυρία Ρέντινγκ, ω συζητήτρια. Και επίση να ευχαριστήσουμε και του συνεισηγητέ. Είναι πολύ σημαντική αυτή η συνεισφορά του Κοινοβουλίου και θα θέλαμε η διαπραγμάτευση να γίνει σε στενή συνεργασία μαζί σας. Όπως γνωρίζετε, το 70% των υπηρεσ... του, το, ΑΕΠ μας προέρχεται από τις υπηρεσίες, αλλά μόνο το 25% των εξαγωγών μας. Η ΤΙΖΑ είναι ένας τρόπος, μια προσπάθεια να αντιμετωπίσουμε την, το πρόβλημα αυτό, την ανισορροπία. Αυτή τη στιγμή, 23 ε, χώρες ε, μέλη του ΠΟΕ συναντώνται για την 16η ε, ε, σειρά, στην, ε, σειρά των διαπραγματεύσεων, συνάντηση σειρά των διαπραγματεύσεων και ελπίζω ότι αυτό θα συνεχιστεί. Είχα τη δυνατότητα να μιλήσω με όλους τους υπουργούς που εκπροσωπούν τις χώρες που θα συμμετάσχουν στην Πίζα στον Ταβός. Ήταν πολύ θετική η ατμόσφαιρα. και επιθυμούν πολλές χώρε να τελειώσουν αυτές τι διαπραγματεύσεις φέτος. Θεωρώ ότι αυτός ο στόχος είναι ρεαλιστικό, αλλά κατά την άποψή μας πιο μεγάλη σημασία έχει το περιεχόμενο παρά η ταχύτητα. Έχουμε λοιπόν πολλή δουλειά μπροστά μας, μεγάλε φιλοδοξίε, και γι' αυτό το λόγο καλωσορίζουμε τις συστάσεις που ε, καταγράφονται στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που θα τεθεί στη ψηφοφορία την Τετάρτη θέλουμε να παρακολουθείτε την διαδικασία των διαπραγματεύσεων. Όπως αναφέρεται, προσπαθούμε μέσω της ΤΙΣΑ να αξιοποιήσουμε ε, τη δυνατότητά μας να, να, να, να ε, εμπορευτούμε υπηρεσίες σε ένα διεθνές περιβάλλον και να μην υπάρχουν πια εμπόδια στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να το κάνουν αυτό. Αυτό αφορά πολλούς τομείς κρίσιμες σημασίες για το Ευρωπαϊκό Εμπόριο Υπηρεσιών. Επίσης, έχει σημασία για εμάς ο πελημερής χαρακτήρας αυτών των διαπραγματεύσεων και αυτή τη συμφωνία. Συμφωνούμε λοιπόν με την αξιολόγησή σα, και εγώ προσωπικά ότι η συμμετοχή στι διαπραγματεύσει και στην ΤΙΖΑ θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν μεγαλύτερη έτσι ώστε τελικά να περάσουμε προ μια συμφωνία πολυμερού χαρακτήρα. Γνωρίζετε ότι αυτή τη στιγμή οι συμμετέχοντες καλύπτουν το 70% του παγκοσμίου εμπορίου υπηρεσιών. Αλλά θα θέραμε να συμμετάσχουν και άλλες αναδυόμενες οικονομίες, ιδίως η Κίνα. Είναι απαραίτητο να δημιουργηθεί μια κρίσιμη μάζα προκειμένου να γίνει πολυμερής κάποια στιγμή συνθήκη. Εμείς προσπαθούμε η δομή και η αρχιτεκτονική μια συμφωνία ΤΙΣΑ να είναι πλήρως συμβατή με τη Γενική ε, Συμφωνία ε, ε, Εμπορίου Υπηρεσιών, την ΚΑΤΣ. Και επίσης θα ήθελα να πω ότι χαίρομαι που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναγνωρίζει τις προσπάθειές μας να γίνει η πραγμάτευση με διαφάνεια και θα προσπαθήσουμε να συνεχίσουμε σε αυτόν τον δρόμο αυτή τη στιγμή τα έγγραφα ε, και άλλες πληροφορίες παρέχονται στην ομάδα παρακολούθησης στο Monitoring Group του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της οποίας προεδρεύει η κυρία Ρέντινγκ. Και εξασφαλίζουμε ότι οι εκθέσεις από όλους τους κύκλους διαπραγμάτευσης δημοσιοποιούνται στο ίντερνετ. Θα ήθελα να απαντήσω σε ορισμένες από τις ανησυχίες που θέτετε στο ψηφισμά σας. Ζητάτε να γίνουν συμφωνίες οριζόντιου χαρακτήρα και ανάμεσα σε αυτές είναι η υποστήριξη των συμφωνιών του Παγκοσμίου Οργανισμού Εργασίας, στην οποία θα πρέπει να συμφωνήσουν όλα τα κράτη. Όμως, για να γίνει πολυμερής κάποια στιγμή στο μέλλον η συμφωνία ΤΙΣΑ θα πρέπει να την βασίσουμε στο GATS, η οποία δεν περιλαμβάνει τέτοιες προβλέψεις. Επομένως δεν θα ήθελα να πάμε τόσο, δεν θα ήταν σκόπιμο να πάμε τόσο μακριά χωρίς αυτό βέβαια να αποκλεί τη δυνατότητα να προσπαθήσουμε τιμερώς να συνεργαστούμε με χώρες ή σε άλλα φόρα να συνεργαστούμε με χώρες ώστε να τις πιέσουμε να ε, υπογράψουν τις συμφωνίες του ILO. Όσον αφορά τώρα τα εργασιακά, τα κοινωνικά και τα πολιτιστικά δικαιώματα, θα εξασφαλίσω ότι θα υπάρχει η δυνατότητα μονομερώς η Ευρωπαϊκή Ένωση να αποφασίσει σε ποιο επίπεδο θέλει να θέσει την προστασία της, κυρίως δεν πρόκειται ποτέ να απεμπολίσουμε το δικαίωμα των ε, περιφερειακών, εθνικών και ευρωπαϊκών αρχών να οργανώνουν την αγορά των υπηρεσιών όπως αυτό περιγράφεται στη Συμφωνία για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό σας διαβεβαιώνω. Τώρα, όσον αφορά τον τρόπο 1, το mode 1, την περιορισμένη απελευθέρωση των υπηρεσιών διασυνοριακά. Εδώ, σε κάποιους τομείς όπως χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, έχουν εκφραστεί ανησυχίες, αλλά άλλες, άλλοι τομείς, όπως για παράδειγμα οι ψηφιακές υπηρεσίες, είναι προς το όφελος της, σε, σε αυτούς τους τομείς είναι προς το όφελος της Ευρωπαϊκής Ένωσης να πάει προς μια απελευθέρωση. Το επίπεδο προστασίας που θέλουμε να διασφαλίσουμε δεν θα τεθεί σε κίνδυνο εξαιτία της ΤΙΖΑ. Επίσης θέλω να επισημάνω ότι οι διαπραγματεύσεις είναι πάρα πολύ δύσκολες. Επομένως, οποιαδήποτε προσπάθεια μετατροπής των ε, standstill θα μπορούσαν να μας ξαναφέρουν στην αρχή των διαπραγματεύσεων. Αλλά σας διαβεβαιώνω ότι αυτό δεν, δεν ε, μας υποχρεώνει σε απελευθέρωση των αγορών πέραν του επίπεδου που θα το επιθυμούσαμε. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί μέλη, ε, θεωρώ ότι το ψήφισμά σα εκφράζει την έντονη υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και μας ζητάτε να συνεχίσουμε τις διαπραγματεύσεις. Είναι ξεκάθαρες ποιε είναι οι κόκκινε γραμμέ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και σας ευχαριστώ γι' αυτό. Σας ευχαριστώ επίσης για τις γνωμοδοτήσει που έχουν εκδώσει σε διάφορες επιτροπές και σα διαβεβαιώνω ότι θα συνεχίσω να συνεργάζομαι στενά μαζί σα. Ευχαριστώ. Ε, Εκ μέρου ε, τη Επιτροπή ε, Απασχόληση και Κοινωνικών Υποθέσεων, ε, το λόγο έχει ο κύριο Χέντελ. Ευχαριστώ πολύ. Είναι πάρα πολύ σημαντικά βεβαίως τα θέματα της ΤΙΖΑ, αλλά τα πιο σημαντικά ζητήματα δεν έχουν αντιμετωπιστεί. Από το 2007 έχουμε 64 υποθέσεις που αντιμετώπισαν με το Ταμείο παγκοσμιοποίηση έναντι της απελευθέρωσης. Γι' αυτό και ζητά η Επιτροπή απασχόληση, η κύριο υλοποίηση και εφαρμογή τουλάχιστον 8 διατάξεων της Παγκόσμιας της Οργάνωσης Εργασίας να ενσωματωθούν στις προτάσεις με τρόπο δεσμευτικό και με συνέπεια κυρώσει επί ε, περίπτωση του. τους. Αυτό όμως δεν το έχει καλύψει η έκθεση. Οι Ηνωμένε Πολιτείε, ε, το Πακιστάν, η Τουρκία δεν φαίνεται να εντυπωσιάζονται από αυτές τις προσπάθειε επίδειξη δυνάμεως. Φαίνεται ότι δεν υπάρχει καμία απόπειρα να συγκρατηθεί η άκρατη απελευθέρωση έτσι ώστε να υπάρχουν ε, συνθήκες έντιμης εργασιακή ανταγωνιστική σχέση. Σας ευχαριστώ εκ μέρους Επιτροπής ε, Ανάπτυξη. Κυρία Σάντσεθ έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Βαλκάρθελ. Θέλω να ευχαριστήσω και όλους όσους ε, εργάζεστε για την χάραξη ε, διαπραγματευτικών γραμμών για να είναι λιγότερο κακή αυτή η συμφωνία, λιγότερο καταστροφική και ε, θέλω να ευχαριστώ κυρίως την κοινωνία των πολιτών που μελέτησαν τα μικρά γράμματα και είδαν πού είναι απαράδεκτη αυτή η συμφωνία της. Όσοι υποστηρίζουν αυτή την συνθήκη φαίνεται ότι με την έκθεση του TTIP τον Ιούνιο έμαθα το μάθημά τους και δεν ήθελα να ξεκινήσω ξεκινήσουμε αυτό το απαράδεκτο κείμενο, αλλά ίσως ε, να ε, προσπαθήσουν να καλύψουν ε, με ωραία λόγια τις πολύ βλαβερές αυτές διατάξεις. Υπάρχει η χρήση των θετικών ε, καταλόγων, ε, έχουμε την απαγόρευση, μάλλον την απόρριψη των ε, ρητρών standstill, της διατήρησης της σα κατάστασης. Σίγουρα δεν θα πρέπει να αναβληθεί η ψηφοφορία λόγω του αριθμού των τροπολογιών, όπως κάποιοι θα ισχυριστούν. Θα πρέπει να ψηφιστούν οι τροπολογίες, γιατί αποδεικνύουν και δείχνουν ποια είναι η βούληση όλων μας εδώ. Ευχαριστώ εκ μέρους της Επιτροπής Οικονομικών Νομισματικών Υποθέσεων το λόγο έχει η κυρία Μόσκα signor presidente onorevoli στόχος ε, ε, της όπως και κάθε εμπορική συμφωνία κατά εμάς θα πρέπει να είναι ε, να παρέχει ωφέλη στους ευρωπαίους πολίτες και εργαζόμενους και καταναλωτές με πρότυπα φιλόδοξα και κανόνες φιλόδοξους που θα ρυθμίζουν ταυτόχρονα βέβαια και την παροχή των διαφόρων υπηρεσιών. Σε ό,τι αφορά τώρα τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, το Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο ζητεί να προωθήσουμε την εφαρμογή και την υλοποίηση διεθνών κανόνων, χωρίς όμως ε, την ανάληψη νέων υποχρεώσεων που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο ε, τους κανόνες που έχει η Ένωση στον τομέα ε, των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Πρέπει να εκμεταλλευτούμε την ευκαιρία που μας δίνει η ΤΙΣΑ για να φροντίσουμε να καταπολεμήσουμε πιο αποτελεσματικά τη φοροαποφυγή, φοροδιαφυγή, τον επιθετικό φορολογικό σχεδιασμό και τα προβλήματα που αφορούν τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες. Ζητούμε επίσης από την Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ε, είναι διαφανής. Έτσι πρέπει να προσεγγίζουμε την ε, κατάσταση για να γνωρίζουν και οι πολίτες τις αποφάσεις ε, που θα ρυθμίσουν την καθημερινότητά τους. Και ελπίζουμε και ολομέλεια να δώσει θετική της ψήφο. Ευχαριστώ. Εξ ονόματος Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, η κυρία Ροζιέρ έχει τώρα το λόγο. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Με τη Συμφωνία για το Εμπόριο και τι Υπηρεσίε έρχεται μια νέα Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών και νέα συζήτηση σχετική στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Συζήτηση η οποία για άλλη μια φορά γύρει τα ίδια ερωτήματα και επισημαίνει τα ίδια προβλήματα που έχουμε δει και σε άλλε συμφωνίε αντίστοιχε. Καταρχά για τη στόχευση. Μια Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών δεν είναι αυτό ο σκοπό, έχει νόημα μόνο εάν ευνοεί τι επιχειρήσει και τον πολίτη τη Ευρώπη. Και αυτό σημαίνει απλέ αρχέ δηλαδή ισότιμος ανταγωνισμός, αμοιβαία πρόσβαση στις αγορές και διατήρηση δυνατότητας για νομοθέτηση προς το ε, δημόσιο συμφέρον. Και επίσης, πολύ συχνά έχουμε το ίδιο πρόβλημα, όπως και εδώ. Δεν υπάρχει διαφάνεια για τους εκπροσώπους, ε, δηλαδή εμάς, εκπροσώπους του Ευρωπαϊκού, των Ευρωπαίων πολιτών, αλλά και για την κοινωνία των πολιτών. Χρειάζεται λοιπόν περισσότερη διαφάνεια Πρέπει να αποφευχθεί η φοροαποφυγή και το κοινωνικό dumping. Θέλουμε να προστατεύονται τα προσωπικά δεδομένα των πολιτών και να αποκλειστούν από την συμφωνία μια σειρά υπηρεσιών, ε, όχι μόνο οι δημόσιε ασφαλώς υπηρεσίες, αλλά και πολιτιστικού χαρακτήρα. Και χαίρομαι που η συγγήτρια έχει δεχθεί κάποιε από τι ε, τροπολογίε αυτέ, που φαντάζομαι ότι την έχουν φέρει αντιμέτωπη και ε, με μέλη τη ομάδα τη γι' αυτό και την ευχαριστώ ιδιαίτερα για την προσπάθεια. Ευχαριστώ. Ρέντ και Επιτροπή Περιφερειακή ανάπτυξη ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Η Δύσα είναι μια ε, βρύτα του πεδίου ε, συμφωνία η οποία θα ε, έχει συνέπειες και στο τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Είναι απαραίτητο λοιπόν να μην στραφεί κατά των κύριων στόχων της πολιτικής της συνοχής που είναι τα κύρια εργαλεία για την πολιτική συνοχής. Δεν πρέπει να ε, κινδυνεύσει η παροχή των υπηρεσιών, όπως λέει και η γνωμοδότησή μας, όπως λέει και η κυρία Ρέντινγκ, η ποιότητα, η ασφάλεια, η ορατότητα, η ε, δυνατότητα υπολογισμού και προβλεψιμότητα είναι απαραίτητη όρη και πρέπει να μην περιοριστεί η δυνατότητα επιλογής για τους Δήμους και τις κοινότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την ΤΙΣΑ. Πρέπει να υλοποιηθούν με αυτόν τον τρόπο μόνο οι στόχοι τη, χωρί δηλαδή να περιοριστούν οι δυνατότητε και τα συμφέροντα των πολιτών. Εάν διαφυλαχθούν, όπω είναι καθήκον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να διαφυλάξει τα συμφέροντα των πολιτών, τότε μπορούμε να έχουμε μια καλή παροχή υπηρεσία. Η γνωμοδότηση τη Επιτροπή των Περιφερειακών τη Περιφερειακή Πολιτική στην έκθεση ΤΙΖΑ. Ο πρόεδρο. Ευχαριστώ. Τον κύριο Άλμπρεχτ δεν τον βλέπω στο έδρανό του. Υποθέτω ότι δεν βρίσκεται στο ημικύκλιο. Επομένως δίνω το λόγο στον κύριο Φαντενκάμπα, εκ μέρους Επιτροπή Μεταφορών. Ευχαριστώ. Η Ευρώπη έχει πολλά προβλήματα. Γνωρίζουμε το πρόβλημα της προσφυγικής κρίσης, της αύξησης του εθνικισμού. Στον τομέα των μεταφορών θεωρούμε ότι υπάρχουν μεγάλες ευκαιρίες που μας δίνει αυτή η συμφωνία. Ας δούμε για παράδειγμα τι θα μπορούσαμε να κάνουμε στον τομέα των σιδηροδρόμων ή των θαλάσσιων μεταφορών. Εδώ υπάρχουν τεράστιες ευκαιρίες για την Ευρώπη. Υπάρχουν επίσης τα κοινωνικά ε, ζητήματα, τα εργατικά ζητήματα που αφορούν τους εργαζόμενους στον τομέα των μεταφερών πολλές φορές αυτοί υποφέρουν από επιρροή που έρχεται εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό που θα ζητούσα λοιπόν από την Επίτροπο και από την κυρία Ρέντινγκ ε, είναι να συνεργαστούν και τους εύχομαι καλή τύχη. Σας ευχαριστούμε. Εκ μέρους της Επιτροπής Βιομηχανίας Έρευνας και Ενέργειας ο κύριος Μπορέλη έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε ως ε, συντάκτης της γνωμοδότησης που υπερψηφίστηκε ομόφωνα στην Επιτροπή Ήτρε. Στηρίζουμε τη γενική αρχιτεκτονική της έκθεσης Ρέντινγκ, ε, ε, διαφάνεια, λογοδοσία, προστασία δημοσίων υπηρεσιών, επίσης κάλυψη των ειδικών αναγκών, ενέργεια, τηλεπικοινωνίες. Θα ήθελα να σας πω στην παρέμβασή μου το εξής. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέλει να συμπληρωθεί η εντολή του Συμβουλίου για να καλυφθούν κάποια λεπτά ζητήματα, κυριαρχία, αμοιβαιότητα, να έχουμε πραγματικά ωφέλη για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Είναι σημαντικό. Πρέπει να διατηρήσουμε το οικονομικό και κοινωνικό μοντέλο της Ευρώπης, αναγνωρίζοντας ε, τη σημασία των δημόσιων υπηρεσιών. Επίσης, έχουμε κάποιες υποχρεώσεις ό,τι αφορά ε, τη διαδικασία πρόσβασης στα έγγραφα, διαβούλευση με όλους τους φορείς ε, λογοδοσία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να ληφθούν υπόψη όλες οι ε, προφυλάξεις, ό,τι ζητούν οι Ευρωπαίοι πολίτες, τους οποίους και κάλωστε εκπροσωπούμε. Θα πρέπει να τους ε, στείλουμε ε, το μήνυμα ότι το Κοινοβούλιο δεν θα ψηφίσει υπέρ μια συμφωνία στην Τετάρτη, αλλά υπέρ μια πιο αυστηρή, συγκεκριμένη εντολή διαπραγματεύσεων. Ευχαριστώ. Κύριο Κάσπαρη έχει τώρα το λόγο. Πρόεδρε, η κυρία Ρέντινγκ έχει οριστεί υποψήφια εκ μέρους της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου ως καλύτερη ευρωβουλευτής της χρονιάς. Επάξια πιστεύω βλέποντας και την έκθεσή της, αλλά ιδιαίτερα θέλω να σημειώσω μια φράση της για την οποία και μόνο θα άξιζε αυτό το βραβείο. Δεν υπάρχει συμφωνία χωρίς προστασία μας είπε. Α, δεν υπάρχει προστασία χωρίς συμφωνία. Ακριβώς αυτό είναι και το μέλημα της πολιτικής μας ομάδας του Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θέλουμε μια συμφωνία καλή, θέλουμε να διαμορφώσουμε τον, ε, την παγκοσμιοποίηση, κανόνες αφής για τον ε, επιχειρηματία, αλλά πάνω απ' όλα για τον εργαζόμενο και τον πολίτη της Ευρώπης. αξιόπιστους κανόνε. Και είναι η δεύτερη φορά τώρα που ασχολούμαστε με το θέμα αυτό ω Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Δεξοδικά. Καλό σημάδι πιστεύω, γιατί στην αρχή των διαπραγματεύσεων το 2013 είχαμε ήδη εκδώσει έκθεση ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τις δικές μας προτάσεις και παρατηρήσεις Η κυρία Ρέντινγκ μαζί με τους συναδέλφους αφιέρωσαν αρκετό χρόνο τους τελευταίους μήνες για να κοιτάξουμε μεγάλη λεπτομέρεια τα πιο σημαντικά για μας σημεία. Και γι' αυτό απευθύνω έκλειση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κυρία Επίτροπε, ενστερνιστείτε τα όσα θα υιοθετήσει την Τετάρτη το Κοινοβούλιο για να σας υποστηρίξουμε με ευρύτατη πλειοψηφία πιστεύω και να έχετε τη μέγιστη δυνατή επιτυχία στη σύναψη αυτής της συμφωνίας για το καλό των πολιτών, για τις καλύτερες υπηρεσίες Γιατί μην ξεχνάμε ότι αν πάει κανεί να κάνει σκίση στο εξωτερικό, χρησιμοποιεί υπηρεσίες στην αλλοδοπή ή παίρνει, αγοράζει μια ασφάλιση ζωή, ένα ασφαλιστήριο ζωή. Είναι το ίδιο πράγμα και έχουν τεράστια σημασία αυτά και για την καθημερινή μα ζωή. Ευχαριστώ. Υπάρχει για κάρτα από τον κύριο για εσά, κύριε Κασπαρή. Δέχεστε την κάρτα, μάλιστα. Ο κύριος Ρόιλε, πρόεδρε, ευχαριστώ. Ρούμπιχ, Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ για την παροχή των υπηρεσιών. Ε, θα φέρει υψηλότερου μισθού, μα λέτε, και ταυτόχρονα θα ενισχύσει την αγοραστική δύναμη. Αν κανεί μπορεί να αγοράζει πιο φθηνά, τότε μπορούν και οι επιχειρήσει μα να γίνουν πιο ανταγωνιστικέ. Πιστεύετε ότι και για την απασχόληση μπορεί να είναι σημαντικό να συνάπτονται τέτοιου είδου συμφωνίε και πιστεύετε ότι μπορούν να υποφεληθούν από τέτοιε συμφωνίε και οι μικρο επιχειρήσει. μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ο κύριος Κάσπαρη απάντηση. Αγαπητέ συναδελφέ, ασφαλώς αυτό είναι ένα από τα πιο σημαντικά σημεία, ότι και θα είναι πιο φθηνές οι υπηρεσίες που θα αγοράζουμε, αλλά και θα είναι καλύτερη η πώληση, η παροχή δηλαδή των υπηρεσιών. Και εδώ ακριβώς πιστεύω ότι έχουμε πολύ καλό ε, ισοζύγιο ω ευρωπαϊκέ χώρε και μπορούμε να βελτιώσουμε ακόμη περισσότερο την παροχή των υπηρεσιών, ταυτόχρονα δημιουργώντα νέε θέσει εργασία. Και αυτό, όπω είπαμε, αφορά όχι τι μεγάλε τόσο, όσο τι μικρέ και μεσαίες επιχειρήσει τη Ευρώπη. Ευχαριστώ. Εμεί ευχαριστούμε κυρία Κίρτον Τάρλινγκ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ την εισηγήτρια και του σκιώδη. Αυτέ οι διαπραγματεύσει είναι γνωστό είναι ότι είναι αμφιλεγόμενες. Οι υπηρεσίε έχουν κρίσιμη σημασία για την οικονομία μα Η ποιότητα των υπηρεσιών έχει τεράστιε επιπτώσει στην, στην κοινωνία, στην απασχόληση κτλ. Όπως γνωρίζετε έχουμε τη δυνατότητα ως κοινοβούλιο να ασκήσουμε βέτο. Εάν το, το κάνουμε αυτό έξυπνα θα έχουμε τη δυνατότητα να οι διαπραγματεύσεις να οδηγήσουν σε κάτι το οποίο θα λειτουργεί για τη δημοκρατία, για τους πολίτες και όχι μόνο για τα κέρδη. Δεν υπάρχει λόγος να δεχτούμε περισσότερο από αυτό που είναι αποδεκτό. Αρχές του Ιανουαρίου στην Επιτροπή Διεθνούς Εμπορέου καταλήξαμε στη συμφωνία η οποία είχε την υποστήριξη της πλειονότητας των πολιτικών ομάδων και θα ήθελα να ζητήσω από όλους τους συναδέλφους να ε, επαναβεβαιώσουν αυτή την εντολή στην Ολομέλεια, δίνοντας τη δυνατότητα στην Επιτροπή μάλλον να μην δώσουν στη δυνατότητα στην Επιτροπή και στα κράτη-μέλη να μας αγνοήσουν, να αγνοήσουν τους πολίτες. Το ζήτημα δεν είναι αν είμαστε υπέρ ή κατά της TTIP. Το ζήτημα είναι να θέσουμε τις κόκκινες γραμμές μας. έχουμε μια συμφωνία η οποία ακολουθεί τους ρόλους ε, και τη λογική της εποχής της αναλογικής ενώ βρισκόμαστε στην ψηφιακή εποχή. Χρειάζεται να επικυρωποιηθούν όλα αυτά. Χρειαζόμαστε νέες ασφαλιστικές δικλείδες. Χρειαζόμαστε να εξασφαλιστεί το δικαίωμα των δημόσιων αρχών να επιβάλλουν κανόνες επιθυμούμε εξαγωγή υπηρεσιών, το οποίο θα δημιουργήσει, λέμε, θέσεις εργασίας στην Ευρώπη, αλλά το ζήτημα επίσης είναι πώς θα δημιουργήσουμε ευκαιρίες στο εσωτερικό, στην αγορά μας, πώς θα εξασφαλίσουμε, πώς θα βεβαιώσουμε μάλλον εκείνους που εργάζονται στον τομέα των υπηρεσιών, ότι είμαστε στο πλευρό του και δεν θα επιτρέψουμε το dumping. Οι κανονιστικές ρυθμίσεις είναι το εργαλείο. Όμως, πρέπει η Κομισιόν να αλλάξει τις προτεραιότητές της στη διαπραγμάτευση. Πρέπει να γίνει ξεκάθαρο στα υπόλοιπα μέρη ότι είμαστε ε, σοβαροί και γι' αυτό το λόγο ζητώ σημαντική υποστήριξη από όλους για αυτό το ψήφισμα στην Ολομέλη. Ευχαριστώ. Κυρία Κίρτον Ντάρλινγκ, υπάρχει γαλάζια κάρτα. Κύριε Ραμινέρ, τη δέχεστε. Ehm, Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. κυρία Κρέτον Ντάρλινγκ θεωρεί ότι είναι πολύ σημαντικά τα συνδικαλιστικά δικαιώματα. Η κυρία Μάλστρομ λέει ότι οι συμβάσεις ε, του Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας δεν έχουν συμπεριληφθεί πλήρως στην Συμφωνία ΤΙΖΑ. Ε, Επομένω, θα επιτρέψει να συμπεριληφθούν κατά την άποψη σας οι διατάξεις των ε, συνθήκων τη Παγκόσμιας Οργάνωσης Εργασία. νέου. Ναι, Απάντηση. Στι διαπραγματεύσει αυτέ, στην ε, συμφωνία GATS σε διεθνέ επίπεδο που θέλουμε να αναθεωρήσουμε, δεν προβλέπεται κοινωνικό κεφάλαιο και δεν συμπεριλαμβάνεται και η κύρωση των προδιαγραφών τη Διεθνού οργάνωση εργασία. Αυτό το ξέρετε πάρα πολύ καλό το συστήσαμε στην Επιτροπή μα και προσπαθούμε να ενσωματώσουμε όρου που θα επιτρέπουν την ε, καταγραφή και των θεμελιωδών εργασιακών δικαιωμάτων στη Σύμβαση στη συμφωνία. Αυτό το έχουμε πει και στην Επιτροπή με μια σαφή απέτηση όλα τα συμβαλόμενα μέρη στη ΤΙΖΑ να κυρώσουν και να υλοποιούν συνθήκες της ILO όχι μέσα από τη συμφωνία αλλά στην πρακτική. Και τελικά η πρακτική είναι αυτό που χρειαζόμαστε και όχι λέξεις ε, πάνω στο χαρτί. Αυτό λοιπόν είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα πρόοδου που διαπιστώνουμε. Ευχαριστώ Μακλάρκιν. Uh, Καλησπέρα. Χαίρομαι κύριε Επιτροπέ που είστε εδώ και σας ε, καλωσορίζω σε αυτή την κρίσιμη σημασία συζήτηση η οποία επηρεάζει δεκάδες εκατομμύρια εργαζόμενους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ΤΙΣΑ θα μας δώσει τη δυνατότητα να αυξηθεί το ΑΕΠ της Ένωσης κατά 206 δισεκατομμύρια, 20 δισεκατομμύρια και δεδομένου ότι το Ηνωμένο Βασίλειο είναι μία από τις μεγαλύτερες εξαγωγούς χώρες υπηρεσιών στον κόσμο, έχουμε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη συμφωνία αυτή. Έχουμε Καταφέραμε στην Επιτροπή να υπάρξει μεγάλη υποστήριξη της έκθεσης, πράγμα που δείχνει ότι πολλοί συνάδελφοι καταλαβαίνουν τη σημασία της ΤΙΣΑ. Από τη μια, πρέπει να φροντίσουμε να είναι φιλόδοξη αυτή η συμφωνία, η οποία να είναι σύγχρονη, να απαντά στα προβλήματα του 21ου αιώνα, όπως για παράδειγμα την εμπορία υπηρεσιών ψηφιακών, αλλά επίσης να βεβαιώσουμε, να εξασφαλίσουμε μάλλον τη συμμετοχή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ταυτόχρονα πρέπει να απαντήσουμε στην ανησυχία του κοινού και των πολιτών. Γι' αυτό έχει συμπληρηληφθεί με βάση την πρόταση της Επιτροπής η προστασία των δημοσίων υπηρεσιών όπως το Εθνικό Σύστημα Υγείας της Αγγλίας έτσι ώστε ε, τα κράτη-μέλη να συνεχίσουν να έχουν το δικαίωμα να προστατεύουν τις δημόσιες υπηρεσίες τους όπως το επιθυμούν. Πιστεύω ότι η έκθεση αυτή μπορεί να έχει την υποστήριξη, υποστήριξη από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να δώσει τη δυνατότητα στην Κομισιό να διαπραγματευτεί με την πίσα με τρόπο που θα ανοίξει ε, ευκαιρίε σε ευρωπαϊκέ επιχειρήσει και τελικά να φτάσουμε και σε μια πολυμερή επικύρωση τη θήκη αυτή. Κύριε Μακλάρκιν, υπάρχει γαλάζια κάρτα από τον κύριο Ντάρμαθ. Δεν τη δέχεστε. Όχι, διότι πρέπει να αποχωρήσω. <laughs> Μα δεν τη δέχεται, κυρία Σχάκε. Μα δεν την έχει δεχθεί. Πρόεδρε, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ηγετική θέση στην εξαγωγή των υπηρεσιών και πιστεύουμε ότι θα έχει ακόμη μεγαλύτερη σημασία αυτό ο τομέα. Οι πάροχοι των υπηρεσιών τη Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολύ ανταγωνιστικοί γιατί έχουμε ένα ανοιχτό περιβάλλον για τι επιχειρήσει. Και έτσι πολλά έχουμε να κερδίσουμε από την ε, αμοιβαία, από το αμοιβαίο άνοιγμα των αγορών διαφόρων χωρών ενώ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άρα την ε, ανταλλαγή ε, παροχής υπηρεσιών σε μεταξύ περισσότερων χωρών. Θα θέλαμε η ΤΙΖΑ να μετατραπεί σε μια πολυμερή συμφωνία και οι υπηρεσίε βεβαίω αναπτύσσονται σε νέου τομεί ταυτόχρονα. Ψηφιακή οικονομία, Φερρυπίν, με ανάγκη να έχουμε πιο ενημερωμένους κανόνες πιο σύγχρονους κανόνες για την παροχή υπηρεσιών και σε τρίτες χώρε η συμφωνία για, τις ε, εμπορικές, ε, για την παροχή εμπορικών υπηρεσιών ε, θα πρέπει ταυτόχρονα όμω να εξασφαλίσει και το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απευθύνει σήμερα με την έκθεσή του στην Επιτροπή την έκκληση να προχωρήσει σε μια φιλόδοξη συμφωνία για τις δημοσιοπηρεσίες μεταφορές, το ηλεκτρονικό εμπόριο, τις οικονομικές υπηρεσίες και τις μεταφορές και ιδιαίτερα θέλουμε να αντιμετωπιστούν τα μελήματα των πολιτών. Θέλουμε να δώσουμε απαντήσεις και να εξηγήσουμε ότι δεν έχουμε λόγο να φοβούμαστε. Το Κοινοβούλιο επικυρώνει φυστάμενη νομοθεσία και προδιαγραφές. Δεν μειώνει το επίπεδο. Θα ακολουθεί τους κανόνες το ελεύθερο εμπόριο. Άρα λοιπόν και στις οπτικοακουστικές υπηρεσίες που έχουμε συμπεριλάβει στην έκθεσή μας για να τις αποκλείσουμε και η ΤΙΖΑ δεν μπορεί να υποχρεώσει κράτη, μέλη και κυβερνήσεις να ανοίξουν μονοπωλιακές σχέσεις όπως αυτές με το νερό ή το ηλεκτρικό ρεύμα. Συμφωνώ λοιπόν με την συγγήτρια και τους σκιώδη συγγητές. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους όσοι συνεργάστηκαν σε αυτές τις πολλές σημαντικές διαπραγματεύσεις και ελπίσουμε ότι θα, θα εξακολουθήσετε να εκπροσωπείτε την Ευρωπαϊκή Ένωση με την παρουσία και την αυτοπεποίθηση που απαιτείται για καλύτερου κανόνε, για εφαρμογή καλύτερα των κανόνων και για όσο δυνατόν μεγαλύτερη συμμετοχή κρατών στη συμφωνία για να είναι και πιο αποτελεσματική. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Σάκε. Υπάρχει η γαλάζια κάρτα από τον κύριο Ντάρμαθ. Τη δέχεστε. Γιατί όχι κύριε Πρόεδρε. Um, uh, Θέλω να ευχαριστώ την κυρία Σχάκε θερμότατα που δέχτηκε τη γαλάζια κάρτα. Έδειξε την ευγένεια που φαίνεται ότι είναι ανήκα να δείξει, το έδειξε τουλάχιστον ξεκάθαρη κυρία Μακλάρκιν. Η ερώτηση είναι η εξή. Πιστεύετε ότι τα εργασιακά δικαιώματα ε, θα πρέπει ύψο φάκτο να περιλαμβάνονται σε όλες τις εμπορικές συμφωνίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή πιστεύετε ότι τα εργασιακά δικαιώματα ορίζονται και αποφασίζονται καλύτερα σε εθνικό επίπεδο απάντηση. Στο ψήφισμα αυτό ε, μιλάμε για τις διαπραγματεύσεις ε, για την ε, Συμφωνία Εμπορίου Υπηρεσιών. Θα θέλαμε σε όλες τις άλλες συμφωνίες να γίνονται σεβαστά τα εργασιακά δικαιώματα όπως αυτά κατοχυρώνονται από τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας. Η συνάδελφός μου πολύ σωστά, κ. Τον Τάλινγκ, λέει ότι είναι πιο σημαντική η πρακτική εφαρμογή των προτύπων και κανόνων και να μην κάνουμε ανεδαφικές ασκήσεις επί χάρτη. Θα πρέπει λοιπόν, λοιπόν και στις ε, συμφωνίες ε, για τις υπηρεσίες να υψώνουμε τον πύχη σε ό,τι αφορά τα πρότυπα και τους κανόνες και σε ό,τι αφορά τα εργασιακά δικαιώματα. Ευχαριστώ πολύ ο Πρόεδρος, κύριο Κούλογλου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ξεκίνησε προσπάθεια προχτές την Παρασκευή από τον Πρόεδρο να αναβληθεί η ψηφοφορία για την Τίζα με διάφορα τεχνικά προσχήματα όπως έγινε και πριν από λίγο καιρό με τη δίδυμη αδελφή της τίζα την DTIP και γιατί ο πρόεδρος θέλει να την αναβάλει γιατί δεν ξέρει αν η ομάδα του θα ψηφίσει υπέρ τη συμφωνία ή κατά. και γιατί δεν το ξέρει γιατί αυτή τη συμφωνία δεν τη χρειάζεται η ευρωπαϊκή ένωση και δεν τη θέλουν πολλοί βουλευτές. υπάρχει ήδη η ΓΚΑΤΣ. αν χρειάζεται αλλαγές ας την εξυγχρονίσουμε. οι μόνοι που προωθούν τέτοιε συμφωνίε είναι οι πολυεθνικές εταιρείε και οι πολιτικοί του εκπρόσωποι. ξέρουμε το έργο απορρίθμιση απορρίθμιση απορρίθμιση των κανόνων και των υπηρεσιών αποδυνάμωση των κρατών να ρυθμίζουν τις υποθέσεις περιορισμός των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων αμφισβήτηση των κανόνων και της ποιότητας εργασίας. ακόμα και τώρα προτείνουμε στο κοινοβούλιο να ζητήσει από την κομισιόν να αποσυρθεί από τις διαπραγματεύσεις όπως έκανε η ουρουάη. ζητάμε εξουσία στις κυβερνήσεις να αλλάζουν πολιτική και συμφωνίες αν αυτό το θέλουν και το ψηφίζουν οι πολίτες. ξεκάθαρη εξαίρεση των δημόσιων υπηρεσιών από την υποσυζήτηση συμφωνία. διαφορετικά υπηρεσίες όπως η υγεία και η εκπαίδευση σε λίγο θα ιδιωτικοποιηθούν. επικύρωση των συμβάσεων εργασίας της διεθνούς οργάνωσης εργασίας προστασία του περιβάλλοντος προστασία των δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής σταματήστε να ψηφίζετε συμφωνίες που υπονομεύουν τα κοινωνικά θεμέλια της ευρώπης. Κυρία Ρέντα, παρακαλώ. Πρόεδρε, ευχαριστώ συνάδελφοι κύριε Επίτροπε. Τα μηνύματα από τους διαπραγματευτές είναι σαφέστατα. Πρέπει να ξαναγυρίζουν στην τράπεζα σχεδιασμού. Δεν καταγράφονται δηλαδή οι απόψει των πολιτών και πάντω όχι του Κοινοβουλίου από τη Συμφωνία. Το δημόσιο συμφέρον δεν έχει ληφθεί υπόψη παρκώ. Οι πολίτες αντιτάσσονται στην ε, απελευθέρωση των δημοσίων υπηρεσιών, θέλουν ρήτρε και άλλα μέτρα που μπορεί να περιορίσουν τα δικαιώματά μας για νομοθέτηση προς το δημόσιο συμφέρον να απαλληφθούν. Και άρα πρέπει να εξασφαλιστεί περισσότερη εμπιστοσύνη. Αυτό το έχει καταφέρει σε έναν βαθμό η έκθεση. Το Κοινοβούλιο είναι η φωνή του λαού σε αυτέ τι διαπραγματεύσει και πρέπει να δείξει μεγαλύτερη υπηρεσία. Πρέπει να απορρίψει ξεκάθαρα και περίφραστα οποιαδήποτε συμφωνία δεν έχει την κατάλληλη προσέγγιση. Πρέπει να είμαστε συνεπεί στι επικρίσει που διατυπώνονται και στην έκθεση και να πετύσουμε την αλλαγή τη εντολή για τη διαπραγμάτευση για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ιδάλω, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να είναι βεβαία ότι είμαστε έτοιμοι και να απορρίψουμε την ΤΙΖΑ. Δεν έχουμε πιστεί ακόμη ότι πρέπει να παραιτηθούμε από την πολυμερή προσέγγιση και να προχωρήσουμε προς ε, πιο εντατικέ συνομιλίε με ορισμένε χώρε, οι οποίε δεν έχουν καν κάτι στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και άρα έχουν άλλα πλεονεκτήματα. Ούτε οι πολίτε συμμετέχουν στη ΤΙΖΑ όπω δεν είχαν την δυνατότητα να φράσουν τι θέσει του και για την TTIP. Και μόνο από διαρροές ενημερωνόμαστε. Πολλά είναι τα σημεία τα οποία μας ανησυχούν. Ενημερωνόμαστε, όπως είπα, από τις ε, διαρροές. Υπάρχουν ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα ε, προσωπικά δεδομένα και την προστασία των καταναλωτών. Χρειάζεται να υπάρχουν ε, πιο σαφείς διατάξεις για την ουδετερότητα του δικτύου, η επιλογή του παρόχου του των διαδικτυακών υπηρεσιών, σημεία στα οποία θα πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση και να μην επιτρέψουμε να απομονωθούμε μέσα σε μια συμφωνία η οποία θα μας επιτρέπει να διαφυλάσσουμε τα ψηφιακά μας δικαιώματα. Ευχαριστώ, η κυρία Μπέγκιν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κυρία Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Συμφωνία για το εμπόριο υπηρεσιών έχει δύο όψεις. Έχει το καλό πρόσωπο, μια αντίστοιχη συμφωνία ανάπτυξη, απασχόληση, προστασία εργαζομένων και από την άλλη πλευρά από τα κείμενα που είδαμε βλέπουμε και μία σκοτεινή ε, πτυχή της ΤΙΖΑ τέλος στις δημόσιες υπηρεσίες όπως τις ξέραμε μέχρι τώρα ή την υγεία ή το σχολείο ή το διαδίκτυο κτλ. κτλ. Τελικά τι από όλα αυτά είναι αυτή η συμφωνία ΤΙΣΑ. Πόρο απέχουμε τη ολοκλήρωση της συμφωνίας, είναι άκρος απόρριτες οι διαπραγματεύσεις και τελικά ποια όψη, ποιο πρόσωπο της συμφωνίας θα επικρατήσει. Εμείς είμαστε εδώ και θα παρακολουθούμε τα πράγματα διότι αργά ή γρήγορα κυρία Επίτροπε θα φτάσει στο Κοινοβούλιο η συμφωνία αυτή την Τετάρτη, την ψηφίσουμε ένα κείμενο κείμενο που θα αναφέρει ξεκάθαρα τις ανησυχίες μας και τις ε, ε, προτάσεις μας. Πρόκειται για την εντολή μας προς τους διαπραγματευτές και ελπίζω να τηρηθούν ε, αυστηρά γιατί θα σας περιμένουμε στη γωνία κύριε Επίτροπε. Κύριε Σομπερμάγη. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Η έκθεση περιλαμβάνει πολλέ υποσχέσει για καλύτερη προστασία των δημοσίων υπηρεσιών, των οικουμενικών υπηρεσιών, ε, και πολλά άλλα αντίστοιχα. Υπάρχει περίπτωση όμως να το πιστέψουν αυτό οι πολίτες. Το έχουμε δει και με την TTIP και από την έκθεση βλέπουμε, διότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί πως έχει κάνει σωστές επιλογές και κάνει υποσχέσεις εδώ και χρόνια ότι τάχα θα προστατευθούν ε, οι δικές μας προδιαγραφές στα των προσωπικών δεδομένων, Φερρυπίν. Η έκθεση ζητεί περισσότερο άνοιγμα σε θέματα για την ελεύθερη διακίνηση των εργαζομένων, Φερρυπίν, ε, σε σχέση με τους ε, ε, εταίρους. Είναι δυνατόν όμως η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει αναλογιστεί τις συνέπειες τέτοιων επιλογών. Συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών και απελευθέρωσης του εμπορίου τέτοιου τύπου μπορεί να οδηγήσουν σε πολύ σημαντικές αλλαγές. Δεν ξέρω αν η εισηγήτρια έχει τόσο στενές σχέσεις όπως ακούγεται με μεγάλους ομίλους όπως η Μπέρτελσμαν, αλλά θα πρέπει να το κοιτάξουμε πιο προσεκτικά. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Επιτίδιος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η συμφωνία για τις ε, συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών ενώ θεωρητικά αποσκοπεί στο να βοηθήσει τις ευρωπαϊκές εταιρείες που παρέχουν αυτές τις υπηρεσίες παγκοσμίω στην πραγματικότητα αποτελεί ένα ακόμη χτύπημα στην ιδέα του εθνικού κράτους. Περιορίζεται ο δημόσιος έλεγχος σε θέματα ε, χρηματοπιστωτικών ε, υπηρεσιών και στην ουσία καταργείται το κρατικό μονοπόλιο σε αυτούς τους τομείς. Το κράτος δεν έχει τη δυνατότητα να παρεμβαίνει για να προστατεύει τα συμφέροντα των πολιτών του και όταν συμμετέχει συμμετέχει σε πολύ μικρό ποσοστό και δεν μπορεί να ορίσει τους κανόνες με τους οποίους ρυθμίζεται η παροχή αυτών των υπηρεσιών. Συνεπώ έχουμε ε, μείωση της ε, κρατική παρεμβάσεω και ε, περιορίζονται και θίγονται τα συμφέροντα τόσο των πολιτών όσο και των μικρών εταιρεών ει βάρο των μεγάλων πολυεθνικών. επιπλέον το κράτο είναι υποχρεωμένο να τηρεί αρχεία αυτών των υπηρεσιών και να ε, παρέχει τα έξοδά του. επιπλέον εάν υιοθετηθούν κάποια στοιχεία τα οποία έχουν προτείνει οι ηπα τότε το κράτο δεν θα μπορεί να δίνει συντάξει στου ε, πολίτε του. κάτι τέτοιο συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην πατρίδα μου την ελλάδα. προσπαθεί να επιβληθεί αυτή η πρακτική τέλος ε, υπάρχει το ενδεχόμενο να έχουμε διαρροή προσωπικών δεδομένων προς χώρες οι οποίες χαρακτηρίζονται από τη μεγάλη διαφθορά τους. Άρα... Ευχαριστούμε. Ο κύριος Βαλές έχει τώρα το λόγο. Η συμφωνία αυτή ανοίγει νέους ορίζοντες ό,τι αφορά την πρόταση στις αγορές, αλλά θα ε, βελτιώσει και τους διεθνούς κανόνες στον τομέα των μεταφορών, των ψηφιακών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, θα καλύπτει και ένα ευρύ φάσμα εμπορικών ε, υπηρεσιών. Είναι προφανές, ε, τουλάχιστον κατά με, ότι πρόκειται για μεγάλη ευκαιρία. Θα έχουμε νέες αγορές για τις μεγάλες επιχειρήσεις, θα μπορέσουμε να εδραιώσουμε τη θέση της Ευρώπης ως ηγέτη στην παροχή υπηρεσιών. Έχουμε στηρίξει μια διαδικασία ισορροπημένη, έχουμε ζητήσει να υπάρξουν πιο φιλόδοξε δεσμεύσει ό,τι αφορά την έρευνα και ε, την τεχνολογία, τι λεπικοινωνίε, μεταφορέ, μεταπιστωτικές υπηρεσίε και άλλου τομεί, Αλλά δεν θα πρέπει να ξεχνάμε και τα δικαιώματα των καταναλωτών. Τέλη περιαγωγή, δηλαδή εισιτήρια, μεταφορές, ε, τα τέλη της χρήσης χάρη στο εξωτερικού κτλ. κτλ. Στηρίζω ε, την εξαίρεση των δημόσιων και των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, των αποκλειστικών υπηρεσιών τη συμφωνία και χαίρομαι που βλέπω ότι στο ψηφιακό τομέα ε, ζητούμε να υπάρξει καθολική απαγόρευση ε, του εντοπισμού των δεδομένων και ζητούμε και την προστασία δεδομένων. Στηρίζω τη συμφωνία. Θέλω να συγχαρώ και να ευχαριστήσω την κυρία Ρέντινγκ για το καταπληκτικό έργο που έχει κάνει μέχρι τώρα. Ευχαριστώ. Σα Σας ευχαριστούμε. Ο κύριος Μάρτιν έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεδομένου, όπως είπαν και άλλοι, ότι το 70% του ΕΠ μας έρχεται από τις υπηρεσίες, είναι δεδομένο ότι η ΤΙΣΑ είναι μια μεγάλη ευκαιρία. Γιατί θα δώσει τη δυνατότητα σε ευρωπαϊκές ε, επιχειρήσεις να δραστηριοποιούν σε μια ενιαία αγορά. Αυτό θα βοηθήσει ιδιαίτερα τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ιδιαίτερα έναντι των μεγαλύτερων επιχειρήσεων. Η ΤΙΣΑ μπορεί επίση να βοηθήσει τους καταναλωτές, ε, επιλύοντας προβλήματα που συχνά έχουν οι καταναλωτές να πρέπει να διαπραγματευτούν με κάποιον πάροχο σε τρίτη χώρα. Επίσης, θα δώσει τη δυνατότητα να προστατευτούν καλύτερα τα δικαιώματα των εργαζομένων. Θα μπορούσε, είπα, και επίτηδε τα είπα όλα υποθετικά. Το κατά πόσον τελικά θα συμβεί αυτό εξαρτάται από το εάν θα προστατευτούν οι δημόσιε υπηρεσίε, το δικαίωμα των κρατών να υποβάλουν κανόνε, εάν θα προστατευτούν τα προσωπικά δεδομένα. Η πολιτική μου ομάδα θα υποστηρίξει την ΤΙΣΑ μόνο εάν τελικά διαπιστώσουμε ότι ανταποκρίνεται στι επιθυμίε μα. Ευχαριστώ. Έχετε μία μπλε κάρτα από τον κύριο Αρνό, κύριε Μάρτιν, τη δέχεστε. Ε, λοιπόν. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μάρτιν και σέβομαι τις θέσεις σας. Αλλά θα ήθελα πολύ συγκεκριμένα κάποιες ακραίες ρήτρε, ιδιαίτερα στο τμήμα 4 των συστάσεων προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπου λέμε ότι δεν δεχόμαστε ακραίες ε, υπερφιλελεύθερες θέσεις. Ε, νομίζετε ότι θα μπορέσετε να υποστηρίξετε μια έκθεση που θα είχε τέτοιες ακραίες φιλελεύθερες ε, ρήτρε. Απάντηση. Και για το θέμα αυτό, όπω και για κάθε εμπορική συμφωνία, δεν, ε, δεν δεχόμαστε ε, ρήτρε, δεχόμαστε το δικαίωμα να ορίζεται μια κυβερνητική πολιτική για την παροχή των δημοσίων υπηρεσιών στο κοινό, όπως πρέπει. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κύριε Πρόεδρε, οι υπηρεσίε είναι σημαντικό τομέα ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Γερμανία ιδιαίτερα. Με όλο και μεγαλύτερη παραγόμενη αξία και μεγαλύτερο μερίδιο στο διεθνέ εμπόριο. Το ακούσαμε και αυτό. Είναι γνωστό ότι το διεθνές εμπόριο γεννά τη δυνατότητα για την εξασφάλιση απόλυτων αλλά και συγκριτικών οικονομικών ε, ωφελών και αυτό βέβαια είναι πολύ σημαντικό, υπογραμμίστηκε ήδη. Η ΤΙΖΑ μπαίνει ως ένα ακόμα λιθάρι στο οικοδόμα του ΠΟΕ εφόσον μπορεί να προχωρήσει θετικά σε μια καλή συμφωνία. Με την έκθεση καταγράφεται ξεκάθαρα η πρόθεση προς διεθνές εμπόριο, σχέσεις εμπορικές ε, διεθνείς, χωρίς όμως να τεθεί σε κίνδυνο η παροχή των οικουμενικών υπηρεσιών. Γι' αυτό και με υπέρ της συμφωνίας και της εντολής. Ευχαριστώ κύριο Σόλτ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, κυρία Ρέντιν, κυρία Συγκεντρία. Η έκθεσή σας συμπεριλαμβάνει μια σειρά από μελήματα, πρέπει να το αναγνωρίσω αυτό και της ε, κοινή γνώμης και των πολιτών. Πολλούς, πολλοί από τους Δήμους, τις κοινότητες έχουν διατυπώσει όμως προτάσεις οι οποίες συμβαστικές σας ε, τροπολογίες δεν έχουν βρει θέση. Έχουν προτείνει παραδείγματι επικοδομητικά να εργαζόμαστε με θετικούς καταλόγους, δηλαδή αυτούς, αποκλειστικούς καταλόγους, αυτούς οι οποίοι αν ε, δεν αναφέρουν κάτι συνεπάγονται πως δεν μπορεί και να καλυφθεί από τη συμφωνία. Πρέπει να ληφθούν υπόψη αυτά και να βελτιωθούν αντίστοιχα οι παράγραφη. Αλλά αγνοήθηκαν οι προτάσεις οι οποίες είχαν σαν στόχο να διαμορφωθούν οι όροι της παγκοσμιοποίησης με σεβασμό στον πολίτη. Πού βρίσκονται λοιπόν οι κόκκινες γραμμές, πού είναι οι όροι των δεσμευτικών διατάξεων που μπορούν να επιβληθούν, κυρία δεν νομίζω ότι μπορούμε να έχουμε την εντολή που θα θέλαμε προς το Συμβούλιο και γι' αυτό δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε την πρόταση. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σήμερα εξετάζουμε το ψήσιμο τη Συμφωνία Τίζα. Μια από τις πολλές ε, συμφωνίες ε, που συζητούνται αυτή την εποχή. Έχουμε τη συμφωνία με τον Καναδά, έχουμε τη συμφωνία TTIP. Σίγουρα ε, πρέπει να, είναι, ε, να λάβουμε υπόψη ότι υπάρχουν θεμητέ ανησυχίε για τι θα συμβεί με τον πλανήτη, το κλίμα κτλ. με τι ανεπιτυχεί ιδιωτικοποιήσει. Καλό το εμπόριο βέβαια, αλλά δεν είναι σημαντικότερο από το περιβάλλον ή από τα δικαιώματα των ανθρώπων. Γι' αυτό και εμεί στέλνουμε στην Κομισιόν ένα σαφές μήνυμα. Το κείμενο έχει καλή διατύπωση σε ό,τι αφορά την προστασία των δεδομένων, την προστασία του δημόσιου τομέα και το καθεξής. Θα μπορούσε όμως να είναι καλύτερο ακόμη. Γι' αυτό και στηρίζουμε τις τροπολογίες των πρασίνων. Είναι σημαντικό να τις υποστηρίξουμε αυτές τις τροπολογίες για να είναι καλύτερες οι διατάξεις για το περιβάλλον, να υπάρξει θετικός κατάλογος και να είναι δυνατή λήψη καλών αποφάσεων και στο μέλλον. Ευχαριστώ πολύ. Για να δω, μάλιστα. Κύριε Άντερσον, ξέρετε υπάρχει γαλάζια κάρτα για εσάς. Τον κύριο Σάν, τη δέχεστε. Παρακαλώ. Πρόεδρε, αγαπητέ συναδελφέ, ε, επικαλεστήκατε τις πράσινες θέσεις και αν καταλαβαίνω καλά θεωρείται ότι δεν λαμβάνονται υπόψη επαρκώ τα οικολογικά μιλήματα. Μια συμφωνία όμως διεθνή για την παροχή των υπηρεσιών δεν μπορεί να γεννά προβλήματα για το περιβάλλον. Ποια είναι τα προβλήματα που εντοπίζετε εσεί, ποια τι σας απασχολεί ακριβώς. Ακούστε, μιλάμε για δημόσιε συμβάσει μεταξύ άλλων. συγγνώμη, συγγνώμη. Λοιπόν, όπω έλεγα, μιλάμε για κανόνε για τι δημόσιε συμβάσει. Για την δυνατότητα λήψεω αποφάσεων ε, που πρέπει να λαμβάνει υπόψη και την αλλαγή του κλίματος. Eh, για τη διαδικασία, παρακαλώ, έχετε ζητήσει εσείς το λόγο. Για διαδικαστικό. Πρόεδρε, κύριος Γκέρικ. Μόλις μάθαμε ότι προκήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τον ιό ΖΙΚΑ η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, είναι έκτακτη είδηση όταν έχουμε να κάνουμε με παγκόσμια κατάσταση ανάγκη Πρόεδρε, πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να προσαρμόσουμε αναλόγω την ημερήσια διάταξη. Αν θέλουμε να είμαστε και παράγον στη, δημο... στο... Στο... στη διεθνή σκηνή και ξέρω ότι δεν ήταν διαδικαστικό. Ίσως να μην ήσασταν στην αρχή της Συνόδου, όμως το αναφέραμε το θέμα. Και νομίζω ότι δείξαμε την αποφασιστικότητά μας. Ε, συνεχίζουμε λοιπόν με τον κύριο Βόικτ. herr präsident werte kolleginnen und kollegen! Äh, πρόεδρε αγαπητοί συνάδελφοι γινόμαστε μάρτυρες σήμερα το απόγευμα για το πώς ο κύριος Βέμπερ πρόεδρος της πολιτικής ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος θέλει όπως δήλωσε στη συζήτηση να προωθήσει με ταχαία ε, άλματα την συμφωνία ΤΙΖΑ και μαζί να εγκρίνουμε όχι μάλιστα να εγκρίνουμε. Ε, θέλει να προωθήσει μια τέτοια συμφωνία την οποία εμείς δεν πρέπει να εγκρίνουμε και μάλιστα με τέτοιες συνθήκες όταν δεν υπάρχουν δηλαδή επαρκείς όροι για την προστασία της οικουμενικής υπηρεσίας για κάθε πολίτη που δεν θα ε, κοιτάει μόνο το κέρδος. Η δημόσια υγεία όταν είναι ιδιωτικοποιημένη δεν μπορεί ποτέ να κοιτάει την υγεία του ανθρώπου. Το ίδιο συμβαίνει και με το ηλεκτρικό ρεύμα όταν ο άνεργος θα μπορεί πια να πληρώνει το λογαριασμό του, ο οποίος θα έχει σε μόνο ε, γνώμονα το κέρδος, θα μένει χωρίς ηλεκτρικό. Οι δημόσιες υποδομές η παροχή της οικουμενικής υπηρεσίας. Είναι ζητήματα μάλιστα τα οποία δεν μπορούν να επαφεθούν στο στα ιδιωτικά χέρια στις επιχειρήσεις δηλαδή οι οποίες επιδιώκουν το κέρδος. Είναι τεράστια η κίνδυνη. Απορρίπτω λοιπόν με την βαθύτατη και την ίδια ακριβώς πεποίθηση με την οποία απορρίπτω την Ευρώπη αυτή των τραπεζών και των κερδοσκόπων. Ο κύριος Φίσας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε. Η έκθεση που συστούμε σήμερα έχει ως στόχο να αξιολογήσει τα, δύο, τα δυόμιση πρώτα χρόνια ε, της εφαρμογής ε, της Συμφωνίας ε, για την παροχή υπηρεσιών και κυρίως για να δώσει κατευθύνσεις προς την Κομισιόν, για να έχει το απαραίτητο απεριθώρια ελιγμό να συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις χωρίς αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να είμαστε σίγουροι για το τι θα γίνει στο μέλλον. Θέλουμε να βοηθήσουμε να υπάρξει μεγαλύτερη διαφάνεια ε, και καλύτερη συνεννόηση μεταξύ των ε, πλευρών στι διαπραγματεύσει. Είναι μια σημαντική συμφωνία για την Ένωση. Είμαστε ο μεγαλύτερο εξαγωγέα υπηρεσιών, 25% παγκόσμιων υπηρεσιών το 2013. Είχαμε εμπορικό πλεόνασμα 170 δις ευρώ στον τομέα αυτό. Επίσης, ε, οι εξαγωγές υπηρεσιών έχουν διπλασιαστεί τα τελευταία δέκα χρόνια. Είναι σημαντικό η συμφωνία να είναι η πλέον πλειονομερής ε, που θα, λαμβάνει, που θα έχει τη δυνατότητα να διαχειρίζεται και να ρυθμίζει προς το γενικό συμφέρον της υπηρεσίας ε, και να εξασφαλίζει τα δικαιώματα των καταναλωτών ε, και την διατήρηση των υψηλών προτύπων και κανόν. Θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Ρέντινγκ για τη δουλειά της. Τα δυόμιση χρόνια των διαπραγματεύσεων διορθών όχι εφαρμογής της συμφωνίας. Ο κύριος Λάγκε, πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Όποιος θέλει να δώσει ένα σύνθημα για αυτή τη συμφωνία θα πρέπει να πει πιστεύω ναι στις ποιοτικέ υπηρεσίες, όχι στο ξεπούλημα της δημόσιας υπηρεσίας. Ναι σε ισότιμες συνθήκες πρόσβαση αγορές και σε πιο ισχυρά εργασιακά δικαιώματα, όχι στο κοινωνικό ντάμπινγκ. Με αυτά τα συνθήματα λοιπόν, αυτές τις λακωνικές φράσεις μπορούμε να περιγράψουμε μια διεθνή συμφωνία για τις ε, υπηρεσίες. Έτσι θα πρέπει να την περιγράφουμε, δηλαδή να αποτελεί μια υγεία βάση ώστε να μην υπάρχει dumping με την απόσπαση εργαζομένων. Και νομίζω ότι η έκθεση πολύ σωστά επισημαίνει τις υφιστάμενες ε, οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η αρχή δηλαδή ότι για την ίδια δουλειά ε, δίδεται ίδια αμοιβή και τα ίδια δικαιώματα για άνδρες και γυναίκες δεν διαταράσσεται. Ιδιαίτερα λοιπόν θέλω να χαιρετήσω αυτή την προσέγγιση και ελπίζω κυρία Επίτροπε η συνεργασία να σημαίνει όχι μόνο ότι δουλεύουμε μαζί αλλά ότι λέμε νέα περίφραστα στο κείμενο ή όχι εάν δεν είναι καλή και είναι μια κακή συμβαστική λύση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Ευχαριστώ. Έχουμε μια περίπτωση όπου το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να παίξει πλήρω το ρόλο του έτσι ώστε να συνδιαμορφώσει την εμπορική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης καταγράφοντας τις διαπραγματευτικές μας γραμμές για την ΤΙΣΑ. Ελπίζω λοιπόν ότι θα γίνει ε, αυτό σε πλαίσιο έτσι, αμοιβαίας συνεργασίας, επικοδομητικό, έτσι ώστε να καλέξουμε σε μια ε, συμφωνία που να και τις ε, χώρες που, όλες τις χώρες που συμμετέχουν, δίνοντας τη δυνατότητα στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να δραστηριοποιηθούν περισσότερο στο εξωτερικό. Είναι μια ευκαιρία για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας, να έχουν ευκολότερη πρόσβαση σε τρίτες χώρες. Κάτι που θα ωφελήσει ε, δεδομένου ότι οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις παρέχουν υψηλής ποιότητας επιχειρήσεις, είναι χρέος μας να δώσουμε αυτές τις επιχειρήσεις, να δώσουμε τη δυνατότητα σε αυτές τις επιχειρήσεις να τις παράσχουν και στις τρίτες χώρες χωρίς εμπόδια. Ευχαριστώ. Κυρία Μινέρ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, η είναι ο μικρός κακός αδελφός ε, της ε, TTIP ε, και της Συμφωνίας των Καναδά και είναι ένας τρόπος να βλέπουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνει ό,τι θέλουν πολυεθνικές και πώς αντιμετωπίζονται οι δημόσιες υπηρεσίες είναι εμφανές. Καλό είναι να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας μας, αλλά η δημοκρατία, τα δικαιώματα των εργαζομένων ε, δεν θα πρέπει να ε, διακινδυνευτούν γιατί αυτό γίνεται με αυτές τις συμφωνίες. Θα υποχρεωθούν χώρες να ανοίξουν ε, τις αγορές τους και ε, θα υπάρξουν κίνδυνοι για τι δημόσιε υπηρεσίε και γενικώ. Έχουμε την τροπολογία 20, όπου ζητούμε από την Κομισιόν να αποσυρθεί από το τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Αν θέλουμε πραγματικά να προστατεύσουμε τι δημόσιε υπηρεσίε. Ε, δεν υπάρχει καλύτερο τρόπο αυτό. Ε, από το να μην δεχθούμε την ΤΙΣΑ. Έχουμε και την τροπολογία 29 και την τροπολογία 49 για την προστασία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Εγώ πιστεύω ότι όπως προβλέπει και το Άρθρο 53 θα πρέπει να τεθεί υπόψη και των Εθνικών Κοινοβουλίων για έγκριση από αυτά η συμφωνία. Και έχουν και τροπολογία 36 που θέλουν να ψηφίσω. Ο κ. Μποβέ έχει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, εδώ και 30 χρόνια προσπαθούν να μας υποχρεώσουν σε, ε, σε μια συμφωνία για την εμπορία των υπηρεσιών. Στον ΠΟΕ δεν είναι δυνατόν γιατί αυτό είναι ενάντια στα συμφέροντα των πολιτών. Και σήμερα άλλη μια φορά φτιάχτηκε ένα μικρό, μια μικρή λέσχη 23 χωρών από τις 190 προσπαθώντας για άλλη μια φορά να υποστηρίξουν και να υποχρεώσουν τον υπόλοιπο πλανήτη να ακολουθήσει τη συμφωνία τους. Κανένα στον κόσμο δεν το θέλει. Και βλέπουμε ότι οι χώρε αρχίζουν να αποχωρούν, ότι το Πεκίνο δεν συμμετέχει. Γιατί? Γιατί αυτή η συμφωνία αντίκειται στο δημόσιο συμφέρον. Είναι κάτι που το γνωρίζουμε εδώ και 30 χρόνια από τις διαδηλώσεις κατά της ΓΚΑΤΣ. Αυτό έλεγαν τότε. Και βλέπουμε με διάφορους τρόπους να, προσπαθούμε, να προσπαθούν να, να επιβληθεί στις διάφορες χώρες μια συμφωνία πολύ χειρότερη από την ΓΚΑΤΣ. Ακόμα περισσότερο προς την κατεύθυνση της απορρίθμισης, της ανοίγματο των αγορών, δεν πρόκειται να προστατευθούν οι δημόσιες υπηρεσίες, οι οποίες έχουν ήδη ε, σε μεγάλο βαθμό απορριθμιστεί. Ο πρόεδρος διακόπτει το μικρόφωνο του μιλήτη. Σας ευχαριστούμε πολύ. Η κυρία Τόμκ. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ το λόγο. Θα ήθελα καταρχάς ε, να ευχαριστήσω την εισηγήτρια κυρία Ρέντινγκ για τις ε, συστάσεις της και να σημειώσω ότι είχα εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος ε, τη γνωμοδότηση στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων. Πολύ δουλειά έχει γίνει στην έκθεση και το γνωρίζω πολύ καλά. Λυπούμε που ορισμένοι θέλουν να ε, παρεμποδίσουν τις διαπραγματεύσεις μια συμφωνία όπως αυτή που θα μπορούσε να οδηγήσει σε μεγάλη ανάπτυξη και νέες θέσεις εργασία στην Ευρώπη. Συχνά διαπιστώνουμε ότι κάποιοι τάσσονται κατά της ε, συμφωνίας, κατά μια συμφωνίας λόγω άγνοιας, γιατί δεν έχουν όλα τα στοιχεία στη διάθεσή τους. Άρα καλό θα ήταν να ε, προβούμε σε μια προσπάθεια ευαισθητοποίηση και ενημέρωση. Άλλοι πάλι αντιστέκονται σε συμφωνίε γιατί θέλουν να διατηρήσουν συνθήκε μονοπωλίου. Ο ανταγωνισμό πρέπει να υπάρχει. Αν δεν υπάρχει ανταγωνισμό όμω, θα υποφέρει ο πολίτη. Ελπίζω λοιπόν να είναι πολύ καλά τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων και ευχαριστώ θερμά για τη συνεργασία. Ευχαριστώ. Ουλσκοκ. Πρόεδρε, εδώ Είμαι Ölskog είναι το όνομά μου. Οι υπηρεσίε, η συμφωνία με την οποία ασχολούμαστε εδώ έχουν να κάνουν περισσότερη ψηφιοποίηση με σαφείς ε, διαχωριστικές γραμμές μεταξύ υπηρεσιών και κανόνων. Δεν μπορούμε όμως να επιτρέψουμε να έχει ε, κοινωνικό ντάμπινγκ, εκμετάλλευση και καταστροφή του περιβάλλοντος ω συνέπεια αυτή η συμφωνία. Χαίρομαι ιδιαίτερω για την απερίφραστη τοποθέτηση του Κοινοβουλίου με την έκθεση η οποία απαιτεί ξεκάθαρα να γίνουν σεβαστές οι κύριες συνθήκες ε, και προδιαγραφέ της διεθνού Οργάνωσης εργασία και καλεί όλα τα συμβαλόμενα μέρη σε κύρωση της, ε, των συνθήκων της ΔΕΕ Οργάνωσης με την προστασία των δημοσίων υπηρεσιών με την εξασφάλιση υπηρεσιών δημοσίου συμφέροντος ε, συμπληρώνεται ένα κείμενο το οποίο ελπίζω ότι θα μπορέσει να ε, τύχει της υποστήριξη από το Κοινοβούλιο για να έχουμε μια καλή διαπραγμάτευση για την ΤΙΖΑ. Ευχαριστώ κυρία κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε. Εκπλήσωμαι από τα λόγια σας. Είπατε στην ομιλία σας ότι το ψήφισμα αυτό επιβεβαιώνει την εντολή μου. Ότι μπορώ δηλαδή να συνεχίσω να διαπραγματεύομαι όπως μέχρι τώρα. Αν όμως ακούσατε τους συναδέλφους μου, τέλος πάντων τους περισσότερους και αν ακούσατε καλά και την εισηγήτρια κυρίως ε, την ε, κυρία Ρέντινγκ, σας είπε ότι ζητεί σαφώ ε, η Κομισιόν να αλλάξει προσανατολισμό και να σεβαστεί κυρίως κάποιες γαλάζιες γραμμές αλλά και κάποιες Κόκκινε γραμμέ. Ποιε είναι οι κόκκινε γραμμέ, σα τι ε, αναφέραμε. Ρητό να εξαιρούνται δημόσιε υπηρεσίε, να μην υπάρχει ε, απελευθέρωση χωρί ε, δυνατότητα επιστροφή, προστασία καταναλωτών, αποουσία κοινωνικού ντάμπινγκ, ε, να σεβόμαστε τα δεδομένα, τα θεμελιώδη δικαιώματα κτλ. Αυτά όμω δεν τα έχετε συμπεριλάβει μέχρι τώρα στι διαπραγματεύσει. άρα το να συνεχίσετε τι διαπραγματεύσει όπω μέχρι σήμερα σημαίνει ότι παίρνετε το ρίσκο στο Κοινοβούλιο η πλειοψηφία να πει όχι στη Συμφωνία των Υπηρεσιών και ζητώ από όλους τους βουλευτές που θα ψηφίζουν αυτό το ψήφισμα να δείξουν συνεκτικότητα και συνέπεια. Δηλαδή αν δεν σεβαστείτε το ψήφισμα να δεσμευτούν ότι θα καταψηφίσουν και τη Συμφωνία. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Ροντρίδια Πινιέρο. Ευχαριστώ, καλώς ήρθατε κύριε Επίτροπε. Εμείς πιστεύουμε ότι είναι πολύ σημαντικό να επικαιροποιηθούν οι παγκόσμιοι κανόνες εμπορίου. Δεν μπορούμε να ρυθμίζουμε το πιο σημαντικότερο μέρος ε, του διεθνούς εμπορίου με παροχημένους ε, κανόνες ε, στην εποχή του διαδικτύου. Θα πρέπει λοιπόν να φρενάρουμε το κοινωνικό τάπ, να εγγυηθούμε την προστασία της ιδιωτικού χαρακτήρα των δεδομένων, να εγγυηθούμε τις επιγραμμικές υπηρεσίες και εμπόριο, τη περιαγωγή, το ίντερνετ είναι στην υπηρεσία των καταναλωτών και βέβαια και μετά και των επιχειρήσεων. Στηρίζω το ψήφισμα διότι θεωρώ ότι καθιστά ξεκάθαρε ε, τι απαιτήσει του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προ την Κομισιόν, έτσι ώστε οι διαπραγματεύσει ε, να ε, οδηγηθούν στη σωστή κατεύθυνση. Θα πρέπει πολύ ξεκάθαρα να είναι σαφέ ότι θα εξαιρούνται όλε οι δημόσιε υπηρεσίε, να γίνονται σεβαστά τα εργασιακά κοινωνικά δικαιώματα των εργαζομένων, να υπάρχει προστασία των δεδομένων, να υπάρχει ρύθμιση ε, για τα χρηματοπιστωτικά και τραπεζικά στοιχεία. Και βέβαια θα πρέπει να γίνεται σεβαστή η πολιτισμική ποικιλομορφία. Πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εσεί ω Επίτροπο που βρίσκεστε εδώ ενώπιον του Κοινοβουλίου απόψε θα πρέπει να έχετε υπόψη σα ε, την άποψη που ε, αποκρισταλώνεται σε αυτό το ψήφισμα, γιατί τελικά την αρμοδιότητα για την διεξαγωγή των διαπραγματεύσεων την έχει μένει η Κομισιόν, αλλά την αρμοδιότητα για απόρριψη ή έγκριση τη συμφωνία την έχει το Κοινοβούλιο. Και εμεί χρειαζόμαστε καλή συμφωνία, αλλά χρειάζεστε προοδευτική και ε, μια συμφωνία που θα σέβεται το, τα, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα ρεσαία δικαιώματα. Αυτή θα ψηφίσουμε ω Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ. Μογέλ. Ευχαριστώ. Η εισηγήτρια κυρία Ρέντινγκ μας είπε πριν λίγο ότι το ερώτημα είναι τι είδους τίσα θέλουμε. Εγώ θα το έθετα διαφορετικά κατά την άποψή μου. Το ερώτημα είναι θέλουμε μια τέτοια συμφωνία, θέλουμε μια τίσα. Και είναι ξεκάθαρο ότι ένα μέρος των μελών του Κοινοβουλίου, καθώς επίσης και ένα μέρος της κοινή γνώμης, διαφωνεί, δεν θέλει καν αυτή, αυτή τη συμφωνία. Γιατί? Γιατί γνωρίζουμε, έχουμε μάθει από το παρελθόν και έχουμε δει πόσο δυσμενείς επιπτώσεις είχαν προηγούμενες παρόμοιες συμφωνίες και η απορρίθμιση της αγοράς. Πρέπει λοιπόν να θέσουμε τα σωστά ερωτήματα. Θα βοηθήσει μήπως είναι κάτι αντίστοιχο με την Directiva Wolkenstein σε παγκοσμίο επίπεδο. Μήπως θα οδηγήσει σε ακόμα περισσότερη απορρίθμιση των χρηματοπιστωτικών αγορών. Εάν η απάντηση είναι ναι, και μας το πει αυτή η Κομισιόν, τότε σίγουρα δεν υποστηρίζουμε αυτήν την ε, συμφωνία, δεν υποστηρίζουμε την διαπραγμάτευση της Επιτροπής, την Επιτροπή ε, να φροντίσει τα συμφέροντα του πολίτη και του εργαζόμενου στην Ευρωπαϊκή Ένωση στη διαπραγματεύση αυτή. Περνάμε τώρα στη διαδικασία Catch the Πολλές ε, αιτήσει έχω, άρα θα δώσω το λόγο με βάση ε, το εξή κριτήριο. Πρώτον, δεν θα μπορέσουν όλοι να λάβουν το λόγο. Επαναλαμβάνω, υπάρχουν πάρα πολλοί που έχουν ζητήσει το λόγο. Όμω, θα δώσω το λόγο σε όλου του εκπροσώπου ε, των πολιτικών ομάδων που έχουν ζητήσει το λόγο και θα δώσω επίση το λόγο σε αυτούς που είτε δεν έχουν μιλήσει ακόμη, είτε έχουν μιλήσει πολύ λίγο. Και σε αυτούς θα δώσω το λόγο. Κατά τρίτον, που θεωρώ και σημαντικό κριτήριο και αυτό, έχουμε δύο ευρωβουλευτές, γυναίκες που έχουν στη στολό και δεν θα τις αφήσω εκτός. Έτσι θα, ξέρω, θα προχωρήσουμε. Ξεκινά η διαδικασία Μπόγκοβιτς. Ε, Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Ο κόσμος αλλάζει ταχύτατα. Διάφορες υπηρεσίες των χώρων των τηλεπικοινωνιών, των μεταφορών και άλλους χώρους αντιστοιχούν σε μεγάλο μερίδιο της παγκόσμια οικονομίας. Ο κόσμος γίνεται όλο και πιο ψηφιακός. Είναι ανωδική η τάση στην παροχή των ψηφιακών υπηρεσιών. Γι' αυτό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να χορηγήσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ένα σαφέστατο ε, εφαλτήριο για τις διαπραγματεύσεις της σε σχέση με τη Συμφωνία ΤΙΣΑ. Η έκθεση της κυρίας ε, Ρέντινγκ είναι ισορροπημένη, προσφέρει ευκαιρίες για την ευρωπαϊκή οικονομία, για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ιδιαίτερα μελήματα εκφράζει για τα δικαιώματα των εργαζομένων, προσπαθεί να απο ε, τρέψει το κοινωνικό ντάμπινγκ, πρέπει να εξασφαλίσουμε καλύτερα δικαιώματα για τον καταναλωτή, γιατί είμαστε όλο και πιο συχνά χρήστες των ε, υπηρεσιών που προσφέρονται σε παγκόσμιο επίπεδο και ασφαλώς πρέπει και το dumping να αντιμετωπιστεί με μεγάλη προσοχή. Πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στις δημόσιες υπηρεσίες που θα προσφέρονται για το δημόσιο και γενικό συμφέρον. Ευχαριστώ. Πιτσούλα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η διαπραγμάτευση που γίνεται αυτή τη στιγμή από 23 μέρη, δηλαδή 50 χώρες, είναι από τις πιο πλέον ευαίσθητες συμφωνίες στον τομέα των πορειτών υπηρεσιών, δεδομένου του μεγάλου αριθμού ανθρώπων που, υποσχολούνται σε αυτό το τομέα και δεδομένου ότι μόνο στο 2013 173 δισεκατομμύρια του ΑΕΠ προήλθαν από αυτόν τον τομέα. Παρά το γεγονό ότι είναι ανταγωνιστικές οι επιχειρήσει Ευρωπαϊκή παροχή υπηρεσιών στον τομέα τη τεχνογνωσία έχουν να αντιμετωπίσουν νομικά εμπόδια. Ταυτόχρονα, η πρόσβαση στην ευρωπαϊκή αγορά είναι περισσότερο εύκολη, είναι πιο απελευθερωμένη, κάτι που δημιουργεί προβλήματα στι μικρομεσαίε επιχειρήσει. Επομένω, τίθεται το ζήτημα τη αμοιβαιότητα, το οποίο πρέπει να, να το συνδυάσουμε με υποστήριξη των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Ζητείτε οι δημόσιες υπηρεσίες όπως η εκπαίδευση και η υγεία να εξαιρεθούν έτσι ώστε οι τοπικές κυβερνήσεις να έχουν τη δυνατότητα να παίξουν το ρόλο τους. Ευχαριστώ. Κύριε Τόμασιτς, ευχαριστώ. Χαιρετίζω τι προτάσει του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για πραγματεύσει συμφωνιών διεθνού επίπεδου. Διότι η δημόσια κοινή γνώμη θεωρεί ότι αυτή η συμφωνία ε, μέχρι τώρα δεν είναι ε, δυνατό να γίνει αποδεχθή... και θεωρούν ότι κάτι τους κρύβουν οι διαπραγματευτέ. Θέλουν διαφάνεια οι πολίτε και επειδή για του πολίτε εμεί ε, δουλεύουμε, πρέπει να απαιτήσουμε διαφάνεια και δημοκρατικό έλεγχο. Σίγουρα ο δημοκρατικό έλεγχο καθιστά πιο πολύπλοκε στι διαπραγματεύσει, αξίζει τον κόπο όμω. Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν και κάποια ζητήματα παράπλευρα θα έλεγα, όπως αυτή η ψύχωση με τη όταν των δύο φίλων, που επιβαρύνουν κάπως ε, τις συζητήσεις. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε να διευθετήσουμε τα πράγματα, όχι κάνοντας μαθήματα ε, στον υπόλοιπο κόσμο, αλλά με τη δημιουργία ενός νομικού πλαισίου που θα δώσει τη δυνατότητα και στις δικές μας μικρομεσίες επιχειρήσεις ε, να τα πολύ ο κύριος Γιάκοφτσίτς. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Καλωσορίζω τι διαπραγματεύσει που θα αναπτύξει εκ μέρου Ευρωπαϊκή Ένωση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρόκειται για ένα εργαλείο πολύτιμο, ένα εργαλείο πολύ σημαντικό όμω που μπορούμε και εμεί με την εντολή να δώσουμε πλευρά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Εάν ε, βεβαίω ε, είναι κατάλληλη η εντολή και αυτό πρέπει να εξασφαλιστεί με την ε, κοινοποίηση του περιεχομένου των διαπραγματεύσεων με τη διαφάνεια. Είναι πολύ σημαντικό ο πολίτης να μπορεί να γνωρίζει και να υιοθετήσει, να υποστηρίξει τα όσα θα αποφασιστούν εδώ. Ιδιαίτερα τα θέματα της περιαγωγής του ηλεκτρονικού εμπορίου, η ανάγκη για προστασία των εργαζομένων, το δικαίωμα μια ε, τοπική αρχή να έχει την επιλογή της περιφερειακής, ε, η περιφερειακά εδρεωμένης υπηρεσίας. Και δεν πρέπει να περιλάβουμε ε, θέματα τα οποία θα οδηγήσουν στην απόρριψη πλευράς των πολιτών της συμφωνίας. Okay, κύριε Αλμπιόλου. Ευχαριστώ πολύ. Τίσα μαζί με τη ΣΕΤΑ και την που είναι μια τριάδα ε, συμφωνιών, όπως τις λένε, ελεύθερων συναλλαγών. Ελεύθερων όμως για να επιβάλλουν τους κανόνες τους πολυεθνικές, ε, ξεπερνώντας κοινοβούλια και δικαστήρια. Ελευθερία ιδιωτικοποίηση των δημόσιων υπηρεσιών. Αυτό σημαίνουν αυτές οι συμφωνίες. Σκλαβιά για τους ε, εργαζόμενους, άνδρες και γυναίκες. Η ΤΙΣΑ θα δώσει τη δυνατότητα στις μεγάλες εταιρείες και ομίλους να διαλέγουν και να καθορίζουν τα εργασιακά δικαιώματα και θα τους δώσει τη δυνατότητα να ε, μεταφέρουν τις υπηρεσίες και τους εργαζομένους ελεύθερα. Θα φέρει τεράστια ανασφάλεια μια τέτοια συμφωνία. Η αριστερά θα ψηφίσει κατά της ιδιωτικοποίησης των δημόσιων υπηρεσιών, κατά της επισφάλειας, κατά της δικτατορίας των πολυεθνικών κυρίες και κύριοι βουλευτές από το ΕΛΚ και από το, τη σασιολιστική ομάδα. Τι θα ψηφίσετε εσείς, γιατί αν ψηφίσετε υπέρ της έκθεσης σημαίνει ότι ψηφίζετε τη συνέχιση ε, των διαπραγματεύσεων ε, για τη ιδιωτικοποίηση επιχειρήσει και για τα δικαιώματα που θα μας κλέψουν. Πρέπει να, πιστε, να ψηφίσετε ναι για τη δημοκρατία και όχι για τι πολυεθνικέ. Ευχαριστώ. Κύριο Ουρτασούν. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Επιτροπέ, το είπε και ο σύντροφο Μποβέ πριν από εμένα. Ε, ξέρουμε τι είδου είναι αυτέ οι συμφωνίε Ό,τι δεν πετυχαίνουμε στον ΠΟΕ, το προτείνουμε μέσω αυτών των συμφωνιών ενισχυμένο. Ξέρουμε ότι έχει έχουν μπλοκαριστεί οι γκάτς και ε, εμείς φοβούμαστε, ε, έχετε κάποιες επιφυλάξεις, ε, δεν μας καθησυχάζετε, μας ανησυχούν οι δημόσιες υπηρεσίες, οι δημόσιες συμβάσεις. Βλέπετε τι γίνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση με την συμφορίες που γίνεται σε επίπεδο δήμων, το 70% του εργατικού δυναμικού που ασχολείται στις υπηρεσίες, μήπως θυγεί. Τελικά μας ανησυχούν όλα αυτά. Πιστεύω λοιπόν ότι πρέπει να στείλουμε ένα σαφές ξεκάθαρο μήνυμα κάνουμε αυτή την εβδομάδα, να το κάνουμε αυτό, ε, αλλιώς να μην υπερψηφίσουμε αυτό το ψήφισμα, γιατί ε, δεν θα δεχθούμε ε, να έχουμε αυτούς τους θετικούς καταλόγους, αυτές τις διαπραγματεύσεις. Είμαστε επίσης υπέρ της διαπραγματευτικής εντολής της Κομισιόν αλλά δεν μας ε, αρέσει αυτό που λέτε ότι εσείς έχετε πάρει το πράσινο φως ε, για τον τρόπο που διαπραγματεύεστε. Αν ίσχυε αυτό δεν θα ήμασταν εδώ σήμερα να καταθέτουμε αυτό το ψήφισμα. Ευχαριστώ. Άρνολ. Uh, Εκεί όπου εκλέγομαι, οι υπηρεσίε έχουν τεράστια σημασία. Γνωρίζετε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο είναι ο μεγαλύτερο εξαγωγό ε, πάροχο υπηρεσιών, ακόμα μεγαλύτερο και από τι Ηνωμένε Πολιτείε. Αυτό είναι ε, στοιχείο από τη στατιστική υπηρεσία της κυβέρνησης μας. Πρέπει λοιπόν να εξασφαλίσουμε ότι τα δικαιώματα του, ε, των 45.000 ανθρώπων που απασχολούνται σε αυτόν τον τομέα θα διασφαλιστούν, τα δικαιώματα του ΗΠΑ θα διασφαλιστούν, αλλά επίσης δεν είναι δυνατόν να κατακτήσεις, να διαγραφούν μονοκονδυλιά εξαιτίας της ΤΙΣΑ. θα δώσει μήπως τη δυνατότητα να αυξηθεί ακόμα περισσότερο η μετανάστευση προς την Ηνωμένο Βασίλειο με όλο και περισσότερου ε, εργαζόμενους. Μήπως θα μειώσει ακόμα περισσότερο τη δυνατότητα των δημοκρατικά εκλεγμένων κυβερνήσεων να τα παρεμβαίνουν. Όλο και περισσότερο λοιπόν ανησυχώ ότι η ΤΙΣΑ θα οδηγήσει προ τέτοιε κατευθύνσεις. Ευχαριστώ το εμπόριο οποιοδήποτε μορφής βασίζεται σε κανόνες. Διαφορετικά ισχύει ο κανόνας της ζούγκλας. Αναφερόμαστε στις δημόσιες υπηρεσίες, αναφερόμαστε στη σημασία της προστασίας των προσωπικών δεδομένων, αναφερόμαστε στη σημασία της αμοιβαιότητας. Αλλά υπάρχει και ένα θεμελιώδης πρόβλημα, θεμελιώδες πρόβλημα που έχει σχέση με τον τρόπο που οργανώθηκαν αυτές οι διαπραγματεύσεις. Εγκρυπτό, με μια εντολή που δεν ήταν ξεκάθαρη και κυρίως επί τη βάση το, που εγκαθίδρυσε τον ΠΟΕ μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ενώ θα έπρεπε αυτές οι διαπραγματεύσεις να γίνονται στο πλαίσιο του ΟΗΕ. Αυτή τη στιγμή γίνονται πίσω από κλειστές πόρτες το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παρεμβαίνει αποσπασματικά και δεν ακούμε τη φωνή των πολιτών. Δεν δίνεται έτσι εμπιστοσύνη στους πολίτες. Δεν σέβεστε έτσι την δημοκρατία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Περνάμε τώρα στην Επίτροπο, την κυρία Άλπστρο, παρακαλώ. Thank you very much, President. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, για τη δυνατότητα να συζητήσουμε αυτή την πολύ σημαντική ε, συμφωνία που διαπραγματευόμαστε η ΤΙΖΑ είναι μια δυνατότητα να εξασφαλιστεί ένα ισότιμο πεδίο ανταγωνισμού για το εμπόριο τη Υπηρεσία με τεράστιο δυναμικό για την οικονομία εν όλο, αλλά και ιδιαίτερα για την Ευρώπη, τη οποία είναι ανοιχτή η οικονομία ε, προ τι επενδύσει, στι επενδύσει απ' έξω, αλλά πρέπει και οι δικέ μα επιχειρήσει να μπορούν να επενδύουν στο εξωτερικό. Χρειάζεται ενημέρωση και επικαιροποίηση συμφωνία ΑΓΚΑΤΣ για να λάβει υπόψη τα νέα δεδομένα της ε, παγκόσμιας οικονομίας και να εξασφαλιστεί και η ασφάλεια δικαίου που πολλοί από σας επικαλεστήκατε. Το ελεύθερο εμπόριο δεν είναι κάτι το καλό από μόνο του, πρέπει να είναι χρήσιμο στη δημιουργία θέσεων εργασίας, επενδύσεων, αλλά και να πλησιώνεται από μια σειρά από ε, κανόνες και ρυθμίσεις. Στόχος λοιπόν είναι να μετατραπεί σε μια πολυμερή συμφωνία η παρούσα διαπραγμάτευση και γι' αυτό συμφωνώ μαζί σας και γι' αυτό προσπαθούμε Διάκα ως το αρχιτεκτόνιμο αυτό να το κάνουμε στο δυνατόν πιο ανοιχτό και περιεκτικό, ώστε να μπορούν και σταδιακά να ενσωματωθούν σε αυτό, ώστε τελικά να καταλήξουμε σε επίπεδο, σε, πλαίσιο ΠΟΕ και άλλες χώρες. Η ΚΑΤΣ δεν προβλέπει υποχρέωση για ε, υπογραφή και κύρωση διατάξεων και συμφωνιών της ΔΟΕ, της Εθνούς Οργάνωσης Εργασίας, αλλά πάντοτε πιέζουμε προς την κατεύθυνση αυτή ως Ευρωπαϊκή Ένωση σε κάθε εμπορική μα συμφωνία προς τις χώρες οι οποίες δεν είναι ενδεχομένω ε, συμβαλόμενα μέρη στη ΔΟΕ. Και συνεχίζουμε να το πράττουμε. Δημόσιες υπηρεσίες, οπτικοακουστικές υπηρεσίες πάντοτε αποκλείονται από την ε, διαπραγμάτευση. Είναι σαφές αυτό και από την εντολή των κρατών μελών και από το όσο είπατε σήμερα, αλλά και σε προηγούμενες ευκαιρίες. Οι υπηρεσίες δημόσιες, όπως η εκπαίδευση, η δημόσια υγεία, η ίδρυψη, ή οπτικοακουστικές υπηρεσίες αποκλείονται, δεν χρειάζεται να ιδιωτικοποιηθούν και αν ιδιωτικοποιηθούν δεν υπάρχει τίποτε στη συμφωνία αυτή, στην TTIP ή σε άλλη συμφωνία που να αποτρέπει μια τοπική ή περιφερειακή ή εθνική αρχή να επανειθνικοποιήσει να την ε, σχετική υπηρεσία, εφόσον αυτό επιλέξει η κυβέρνηση. Επίσης ε, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα ως προς την ισότιμη πρόσβαση, την προστασία των ε, προδιαγραφών δημόσιας υγείας του περιβάλλοντος. Μπορούν να εισάγουν, να εισάγουν τέτοιες διατάξεις όπως το επιθυμούν οι αρχές. Προσπαθούμε να συμβάλλουμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση στη διαφάνεια, εμπιστος από τις προτάσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και η συνοπτική περιγραφή των διαπραγματεύσεων είναι διαδικτυακά διαθέσιμη. Εσείς ως Ευρωβουλευτές έχετε πρόσβαση σε κάθε έγγραφο, αλλά βέβαια πρόκειται για μια διαπραγμάτευση στην οποία συνεχίσουμε και με άλλες 22 χώρες. Δεν μπορούμε δηλαδή δεν μας επιτρέπεται νομικά να δημοσιεύσουμε τις προτάσεις του Περού, της Νέας Ζηλανδίας, της Αυστραλίας, Τουρκίας, του Πακιστάν πρέπει να είναι δική τους η απόφαση. Λυπούμε που δεν επέλεξαν το δρόμο της διαφάνειας όπως εμείς, αλλά εμείς δεν μπορούμε να δημοσιοποιήσουμε, να δημοσιεύσουμε τα δικά τους έγγραφα. Γι' αυτό πολλές φορές ε, προτάσεις και σχέδια ακόμη προτάσεων χωρών διαραίουν μέσω του τύπου, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είναι τελικές αποφάσεις, είναι μόνο σχέδια προτάσεων προς χωρών και πολλοί από εσά ε, το επισημάνατε. Έχουμε αμέσω μερικές φορές απορρίψει κάποιε από τις προτάσεις αυτές, αν δεν είναι κατάλληλε. Πάντως εμείς πιέζουμε προς τη διαφάνεια, ώστε το δυνατόν περισσότερο όπω ε, λέτε και εσείς. στο τέλος της διαδικασίας και εσείς όπως και τα κράτη-μέλη θα τοποθετηθείτε ασφαλώς. Διαπραγματευόμαστε για την ΤΙΣΑ με βάση εντολή που μας έχουν χορηγήσει 28 κράτη-μέλη. Έχετε και εσείς τοποθετηθεί κατά την εκκίνηση των εργασιών. Βεβαίως ε, λαμβάνω υπόψη τα μελήματα που εκφράσατε, τα ε, σημειώνουμε και θα συνεχίσουμε να τα λαμβάνουμε υπόψη, όπως άλλωστε και τα μελήματα που έχουν εκφραστεί και εκτός της ε, του ημικυκλίου. Αλλά ταυτόχρονα δεν πρέπει να λησμονούμε ότι είναι τεράστια ενεργεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι υπάρχουν εκατομμύρια ανέργων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η ΤΙΖΑ, όπω και άλλε εμπορικέ ε, συμφωνίε, είναι ο τρόπο να εξασφαλιστούν και οι θέσει εργασία και η ανάπτυξη ε, και οι επενδύσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπω θέλουμε. Άρα πρέπει να βρούμε τη χρυσή τομή. Χαίρομαι για την υποστήριξη που προσφέρετε με το ψήφισμα. Θα συνεχίσουμε, όπω είπαμε, τι διαπραγματεύσει. Αυτή τη στιγμή είναι να εξελίξει ένα γύρο διαπραγματεύσεων αυτή την εβδομάδα ακόμα και βεβαίω θα σα ενημερώσουμε μόλι ολοκληρωθεί και ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε μια συμφωνία που θα επιτυγχάνει αυτή η χρυσή τομή που έχετε ζητήσει και βεβαίω πολύ ευχαριστώ. Θα συνεχίσουμε την επαφή και την επικοινωνία. Κυρία Ρέντινγκ, ευχαριστώ για την καταπληκτική αυτή υποστήριξη και τη μεγάλη πλειοψηφία που έχετε εξασφαλίσει, όπω βεβαίω και τι άλλε επιτροπέ με τι νομοδοτήσει του και του χιώδει Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε και τώρα κυρία Ρέτιν για δύο λεπτά εισηγήτρια. Κύριε Πρόεδρε, όπως ε, φάνηκε από τις ε, περισσότερες τοποθετήσεις, ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει συμπήξει ένα ενιαίο μέτωπο και ζητά πλήρη διαφάνεια. Πιο δίκαιους εμπορικούς κανόνες αμοιβαιότητες αγορές, δικαίωμα ρύθμισης προστασίας και περισσότερα δικαιώματα για τους καταναλωτές. Σημαντικότερε πολιτικές ομάδες ε, παίρνουν την κατάσταση στα χέρια του προ αυτή την κατεύθυνση. Η παγκοσμιοποίηση και η ψηφιοποίηση των οικονομιών μας ε, είναι γεγονό. Το ερώτημα λοιπόν το εξή. Θέλουμε η Ευρώπη να είναι μία αδασμολόγητη ήπειρος, αλλά να μην υπάρχει ούτε πίστοτε νόμος. Νομίζω ότι θα πρέπει να είναι η απάντηση του Κοινοβουλίου. Όχι, θέλουμε να συγγράψουμε σήμερα τους κανόνες του παιχνιδιού για να μην τους υποστούμε αύριο. Ε, θέλουμε μια συμφωνία που θα προστατεύει τις επιχειρήσεις μας, που θα προστατεύει τους συμπολίτες μας και ναι, θέλουμε μια αλλαγή πολιτικής μετά τις ευρωεκλογέ του 2014 ε, μια νέα πνοή ε, έχουν πάρει οι εμπορικές συμφωνίες και εμείς θέλουμε ε, να υψώσουμε το λάβαρο. Εάν οι συστάσεις μας τηρηθούν θα βοηθήσει για περισσότερη ανταγωνιστικότητα για τις επιχειρήσεις, θα υπάρξει ένα δίκτυο ασφαλής για τους πολίτες, Γι' αυτό λοιπόν απευθύνω έκκληση στους ε, πολιτικούς και στις διάφορες ομάδες να διατηρήσουν την ε, ισχυρή υποστήριξη που μας έδειξαν γιατί μόνο με μεγάλη πλειοψηφία στην Ολομέλεια θα ληφθούν υπόψη ε, τα αιτήματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όπως είπε ο πρόεδρος της Επιτροπής Ίντα στα γερμανικά. Ένα σαφές ναι στο κείμενο, ένα σαφές όχι σε μια σαθρή σε ένα σταθρό συμβασμό. Ευχαριστώ πολύ